Το Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η δήλωση του ε, ε, Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επί των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2012. Και καλωσορίζω βέβαια τους προσελθόντες και θα λάβει τον λόγο ο πρόεδρος του Συμβουλίου κύριος Φανρόμποϊ. Παρακαλώ κύριε Φανρόμποϊ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από την σύντομη αλλά ε, καλοδεχούμενη και συγκινητική απονομή ε, του ε, βραβείου Νόμπελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγμα το οποίο θεωρήθηκε ως ε, σωστή αποτίμηση του έργου μας κατά το παρελθόν είναι μια πρόκληση να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας στο μέλλον επικεντρωνόμενοι στα κυριότερα θέματα για την υλοποίηση της ε, ε, εμβάθυνσης ε, της Οικονομικής Ένωσης και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης δαπανίσαμε χρόνο για ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής το οποίο αφορά την πλήρωση της ε, χειρεύουσας έδρας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας, πράγμα το οποίο θίγει και από μένα και από τον Πρόεδρό σας στην παρέμβασή του κατά την έναρξη αυτής της συνεδρίασης. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προαχθεί η ισότητα γυναικών και ανδρών είναι ένας στόχος ο οποίος ε, καθορίζεται και συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη. Εχθές με την ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή α, εκφράζεται <clears throat> μια κατανοητή ε, ανησυχία ότι πολλά πρέπει ακόμα να επιτευχθούν ιδιαίτερα όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά επίσης ε, σημειώνουμε και την παρατήρηση της Επιτροπής ότι τα προσόντα, επαγγελματικά προσόντα του υποψηφίου με κανένα τρόπο δεν αμφισβητούνται. Από πλευράς μου στην ε, προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απίθυνα ένα στεναρό αίτημα, μια έκκληση στους αρχηγούς καθώ και κυβερνήσεων να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν και υποψηφίου για τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ε, στην ενθάρρυνση αυτής της διαδικασίας ενεργά. Ελπίζω ότι με την νέα αυτή δέσμευση για την ισορροπία των φύλων το Κοινοβούλιο θα βασίσει την τελική απόφαση επί του σημερινού υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποκλειστικό κριτήριο τα επαγγελματικά του προσόντα διότι πραγματικά επήγει η πλήρωση της ε, χειρεύουσας αυτής θέσης. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι ας περάσουμε στα οικονομικά θέματα τα οποία βρισκόντουσαν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας. Πρώτα απ' όλα ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης συνεχίζουμε να υφιστάμεθα τα πλήγματα από την έλλειψη ανάπτυξης. 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα οι νέοι πλήττονται από την ανεργία. Συνολικά οι προβλέψεις για το επόμενο έτος είναι πολύ μετριοπαθείς. Επόδεινα συνειδητοποιούμε το ποιες ε, επιπτώσεις έχει αυτή η κατάσταση στις κοινωνίες μας. Σε αρκετές χώρες οι προσαρμογές είναι πολύ, πιο, ε, είναι πολύ δρυμύτερες και παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι ε, αναμέναμε. Τώρα, η εξυγίανση των ελλημάτων και η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας θα ήταν αναγκαία στοιχεία και χωρίς την κρίση που διανύει τώρα οικονομικά η Ευρωζώνη. Γι' αυτό είναι τόσο περισσότερο αναγκαίο να επιμερίσουμε τα βάρη αυτής της προσαρμογής με δίκαιο τρόπο όσον αφορά τις πολιτικές που θα στοχεύουν στην μείωση και αντιμετώπιση της ε, ανεργίας. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα εργαλεία και μέσα της πρέπει να ε, δράσει και να συνδέσει συνδράμει όσους χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προώθηση των κοινωνικών στόχων σε μια ανάπτυξη πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και ο ίστατος στόχος μας. Οι δεσμεύσει υπό το Σύμφωνο Σταθερότητα, ε, Ανάπτυξης και δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης δεν μπορούν οι δεσμεύσει αυτές να αναμείνουν περισσότερο. Πρέπει να προχωρήσουμε με δραστήριο, με δραστήριο τρόπο και να μεταφράσουμε τις δράσει μας με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι επίσης αναγκαίο να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε μέτρα για την ε, κοινωνική ολοκλήρωση, λαμβάνοντα υπόψη την ε, προαγωγή τη ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα ε, και την ενδυνάμωση του διεθνού εμπορίου. Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο θα συζητήσουμε το πολιετέ οικονομικό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό, προϋπολογισμό που θα στοχεύει στην ανάπτυξη. Παρότι είναι λιγότερο από το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, θα πρέπει να είναι ένας επενδυτικός προϋπολογισμός που θα έχει τεράστια επίπτωση στην ανάπτυξη. Φυσικά η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη είναι ένα στοιχείο που έχει σημασία ιδιαίτερη για το να μπορέσει η εσωτερική ζήτηση να τονωθεί. Επ' αυτού τώρα έχουμε τα πρώτα, ε, την πρώτη ε, συλλογή στοιχείων σωρευτικά. Σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε τα αποκαλούμενα spreads που μειώνονται σημαντικά σε σχεδόν όλες τις ε, χώρες της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο στις περισσότερες χώρες. Η, η ε, δημιουργία και προώθηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Εποπτείας είναι ένα σημαντικό μέτρο και έχουμε προωθήσει αυτό το στόχο ώστε να βρίσκεται ε, στο ύψος των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ η δημιουργία του μηχανισμού ασφαλείας. Ε, έχουμε και την ε, ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας όπου συγκεκριμένη σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης καλωσόρισαν το στένος Ευρωπαϊκής της ελληνικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να επενέθηκαν οι προσπάθειες που έγιναν. Η ε, ο Ευρωομάδα θα συζητήσει και θα εξετάσει αυτή την πρόοδο υπό το φως της έκθεσης της Τρόικας και υπό το φως της συνεργασίας αυτής η ε, Ευρωομάδα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ε, ομάδα των τεσσάρων προέδρων επίσης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Και από πλευρά ε, του ε, γραφείου μου και η συνεισφορά σε σχέση με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αντιπροσωπεία του, η συνεισφορά ήταν πολύ σημαντική. Συνάντησα και κάποιους από τους εισηγητές σας, προέδρους επιτροπών. Αυτή ήταν μια ενδιάμεση έκθεση που στόχευε στο να αποσαφηνίσει τις, τους και τις κατευθύνσει. Ε, και το επίπεδο υποστήριξης για διάφορες ιδέες ε, που απέρευσαν όσον αφορά τις, ε, τα συμπεράσματα <clears throat> του Δεκεμβρίου. Επικεντρωνόταν στην προσπάθεια που έπρεπε να επιτευχθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή να συνεχιστεί αυτό το έργο και πρότεινε ένα συγκεκριμένο χρονοπλαίσιο και ένα οδικό χάρτη που θα υποβληθεί κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ώστε να μπορέσουν όλα τα στοιχεία να δημιουργηθούν επί των οποίων θα βασίζεται η ένα πραγματικό EMU. Η άμεση προτεραιότητά μας ήταν η οικονομική ολοκλήρωση. Τον Ιούνιο συμφωνήσαμε να, να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζών και ε, ε, η κρατική υπερχρέωσης. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού SSM, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μην υπάρξει περαιτέρω μόλυνση. Και γι' αυτό μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 θα πρέπει να έχει υπάρξει τελική ε, λειτουργική συμφωνία. Όταν θα, έχει, όταν θα μπορέσει αυτό να επιτευχθεί θα μπορέσουμε άμεσα να δραστηριοποιηθούμε. Έχουμε τεράστια ευθύνη που επομιζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το φιλόδοξο χρονορίζοντα. Δεν μπορούμε να ε, υποστούμε τον κίνδυνο να ε, χάσουμε την αναγκαία αυτή όθηση. Θα πρέπει για το, την εποπτεία αυτή να υπάρξει η εξής διαφοροποίηση. Πρέπει να υπάρξει σαφής ε, νομισματική, ε, νομισματική, ε, νομισματικός επιμερισμός ευθυνών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εποπτικές δραστηριότητές της. Θα πρέπει οι εθνικές αρχές να μπορούν να εμπλέκονται στο εποπτικό έργο και στον σχεδιασμό για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και τέλος, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι πλήρης και διαφανής. Όλα τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα και προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Αυτός ο ανοιχτός χαρακτήρας θα πρέπει να αντανακλάται και στην ε, διοικητική δομή με τις ε, αναγκαίες ε, υποχρεώσεις και δικαιώματα από πλευράς όλων. Το SSM είναι ένα πρώτο θεμελιώδες βήμα προς ένα πλήρες πλαίσιο στον ε, χρηματοοικονομικό τομέα. Άλλα βήματα θα πρέπει να γίνουν και μάλιστα γοργά. Ε, ξεκινώντας με τον εναρμονισμό των ε, εθνικών προγραμμάτων όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει έναν ενιαίο μηχανισμό. Όπως συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, άμεσος, άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης θα είναι φυκτή εφόσον το SSM θα έχει αρχίσει να λειτουργήσει λειτουργεί θα έχει εγκριθεί. Ζητούμε από την Ευρωομάδα να συντάξει τα αναγκαία κριτήρια. Για ένα σταθερό οικονομικό και νομισματικό πλαίσιο χρειαζόμαστε η ενισχυμένα πλαίσια για τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά. Ήδη έχουν γίνει πολλά επ' αυτών. Να το διατυπώσω ως εξής. Αν χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλα τα μέσα που έχουμε την εξαπλή πρόταση, την ε, ε, επερχόμενη διτή πρόταση, ΠΑΚ, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τις συστάσεις συγκεκριμένα για τα επιμέρους κράτη-μέλη, χρησιμοποιώντας ε, το μηχανισμό ε, σταθεροποίησης και αποκατάστασης ανισοτήτων, τότε θα έχουμε κάνει ό,τι είναι αναγκαίο. Όμως, για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμα των προοπτικών, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποσβέσουμε τα οικονομικά πλήγματα και τις αποκλήσεις. Εδώ κάποιες νέες σκέψεις στην έκθεσή μου ε, έτυχαν προσοχής. Από κοινού με τους συναδέλφους ε, λάβαμε την εντολή να εξετάσουμε επ' αυτόν το τι μπορεί να γίνει μεταξύ της σήμερα και του Δεκεμβρίου. Μία από αυτές τις προτάσεις είναι ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ατομικές συμφωνίες ε, συμβατικού χαρακτήρα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ανταποκρινόμενα στις συστάσεις για την προώθηση της απασχόλησης και των θέσεων απασχόλησης. Ε, μία άλλη δυνατότητα είναι το οικονομικό δυναμικό ε, και αυτή η ιδέα θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και συμφωνήθηκε ότι αυτό δεν συνδέεται, δεν συνδέεται, το τονίζω αυτό, σε σχέση με την ε, ε, προετοιμασία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα είναι κέρια σημασία στο καινούριο EMU να είναι πλήρως ε, ε, νομιμοποιημένο και να διασφαλίζεται η λογοδότηση και ως γενική αρχή θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο δημοκρατικός έλεγχος θα πρέπει να διασφαλίζεται στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στο ε, νομικό πλαίσιο και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την, εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης της Ένωσης. Επίσης όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική επικεντρωνόμαστε σε δύο κύρια θέματα. Πρώτον, τις σχέσεις μας με την Κίνα κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν και βλέποντας και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ε, σε σχέση με την σύνοδο του Σεπτεμβρίου με την Κίνα έχουμε μια θετική προοπτική. Όπως γνωρίζετε γίνεται αυτή τη στιγμή η αλλαγή ηγεσία όπως συμβαίνει μια φορά κάθε δεκαετία εκεί. Η ανταλλαγή απόψεων με τους Κινέζους πρέπει να διασφαλίζει ένα επικοδομητικό πλαίσιο σε σχέση με τη νέα ηγεσία. Θα πρέπει τα μηνύματά μας προς το Πεκίνο να περάσουν ε, με τον εύθετο τρόπο και, ε, ε, και τα σημαντικά δυσκολότερα μηνύματα επίσης. Θα έχουμε λοιπόν έτσι μια μακρο, πιο μακροχρόνια προοπτική. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα προετοιμάζοντας την επόμενη σύνοδο που θα διαξαρθεί στην Κίνα το φθινόπωρο, το, με συγχωρείτε την άνοιξη του 2013. Δεύτερον, σε σχέση με τις περιοχές κρίσεων στην παγκόσμια σκηνή Συρία, Ιράν και Μαλή. Η κατάσταση αφορούσε την ασφάλεια την ανθρωπιστική, ε, τις ανθρωπιστικές ανάγκες και τις περιφερειακές επιπτώσεις στην υπομεσημβρινή ε, Αφρική, υποσαχάρια Αφρική Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί αποφασίσαμε να επιταχύνουμε το σχεδιασμό μας για μια πιθανή εμπλοκή σε στρατιωτικό επίπεδο για τη διαχείριση της κρίσης εκεί και την υποστήριξη μιας διεθνούς ένοπλης δύναμης σύμφωνα με το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2071. Ολοκληρώνω, ήταν μια θετική σύνοδος, καλή για την Ευρώπη και θα υπάρξει ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που θα μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 2013. Τώρα, μεταξύ της σημερινής ημερομηνία και του Δεκεμβρίου θα συνεχίσουμε την εργασία μας για να ενισχυθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είναι η πιο σημαντική συνεισφορά για την ανάπτυξη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα λάβει τον λόγο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαρόζο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, αγαπητά μέλη. Η προηγούμενη συνάντηση του Συμβουλίου ήταν η τρίτη αυτό το φθινόπωρο για να καταλήξουμε σε αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους στόχους μας. Πρώτον θα πρέπει να προχωρήσουμε με τη συμφωνία του Ιουνίου ε, βλέπουμε ότι η κρίση παραμένει, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν πλέον την οικονομική ύφεση, η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή και θα υπονομεύσει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή και συνειδητοποιώ την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Η εφαρμογή του συμφώνου λοιπόν είναι κάτι πραγματικά το πάρα πολύ σημαντικό ε, και είναι θέμα αν θέλετε επιδίωξης της δικαιοσύνης και της ισότητας. Σε πολλές χώρες οι πολίτες κάνουν τεράστιες θυσίες για καταστάσεις που δημιουργήθηκαν λόγω του υπερβολικού δημοσίου χρέους στον δημόσιο τομέα αλλά και της ανεύθυνης συμπεριφοράς τμήματων του ιδιωτικού τομέα. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε λοιπόν τρόπους να ενισχύσουμε την ελπίδα, την ανάπτυξη και να υπογραμμίσουμε τις προσπάθειες που κάνει η κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις για το σύμφωνο αυτό ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι ότι το σύμφωνο αυτό και το πολύ μεγάλο πακέτο επενδύσεων, σχεδόν 100 ε, δις ευρώ, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Κάποια πρώτα βήματα έχουν γίνει, αλλά όχι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή προσυζήτηση, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και ε, καιρός είναι οι προτάσεις αυτές να γίνουν πραγματικότητα. Ίσως εδώ να δώσω κάποια παραδείγματα. Τους επόμενους δύο μήνες θα πρέπει να γίνουν κάποιες συμφωνίες για τα venture capital ε, και θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες προτάσεις οι οποίες θα ορίσουν με σωστότερο τρόπο τη λειτουργία αυτών των αγορών. Ε, ο φόρος στην αποταμίευση σαν παράδειγμα, οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, ε, τα επαγγελματικά προσόντα Όλα αυτά είναι διαφορετικοί τομεί, προ του οποίους θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο. Πρέπει να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις να θέσουν σε λειτουργία τι συμφωνίε του Μηνό Ιουνίου. Έτσι και εμείς από πλευράς μας θα μπορέσουμε να περάσουμε στην τελική φάση διαμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη είναι σαφές ότι και ο χρηματοοικονομικός τομέας πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Η τελευταία απόφαση για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για μια απόφαση του Συμβουλίου που να επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα και θα παρουσιάσουμε παράλληλα και ένα πρόγραμμα δράσης ε, για τις ε, απάτες στον τομέα της φορολογίας και για τους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Η Επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να εισάγει και ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για την νεότητα έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες αυτών που εγκαταλείπουν την επίσημη εκπαιδευτική θα έλεγα πορεία μέσω προτάσεων κατάρτισης επαγγελματικής και εξειδικευμένη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ποιοτικό πλαίσιο για την επαγγελματική κατάρτιση, βελτιώνοντας τις δυνατότητες των νέων να προχωρήσουν σε έβρεση θέσεων εργασίας. Αγαπητά μέλη, δεν είναι μόνο το σύμφωνο αυτό σταθερότητας και ανάπτυξης το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να υπάρξει και απόλυτη συμφωνία για τον μηχανισμό εποπτείας των πιστοτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγοντας σε μια συμφωνία πάνω σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ε, σε σχέση με την ικανότητά της να λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις σε περιπτώσεις κρίσης. Ας μην αγνοήσουμε λοιπόν αυτή την, ε, αυτό το δύσκολο θέμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση θα έλεγα αν θέλουμε πράγματι να ενισχύσουμε την νομισματική και οικονομική ένωση. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στις διαπραγματεύσεις, ε, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε πολλές από τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει δηλαδή να είναι ανοιχτή αυτή η εποπτική αρχή σε όλες τις χώρες που θέλουν να συμμετέχουν δεν χρειαζόμαστε εμείς ακόμα περισσότερες διαιρέσεις ανάμεσα στην Ευρωζώνη και τα υπόλοιπα μέλη. Απαιτείται επίσης να υπάρξει σωστή ανάληψη ευθύνης για τις δραστηριότητες στο επίπεδο όπου αναλαμβάνεται και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να φύγει τον ενιαίο χαρακτήρα της ε, ενιαίας αγοράς, τον χαρακτήρα της ενιαίας αγοράς και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παρεμβαίνει κανείς σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ευρωζώνη στα πλαίσια αυτής της ε, εποπτείας. Σε όλους αυτούς τους τομείς λοιπόν συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν για την Τραπεζική Ένωση μέχρι το τέλος του χρόνου και ελπίζω όλα τα μέλη να σεβαστούν την ανηλυμένη τους υποχρέωση να μην ξεχνάμε γιατί εμείς προχωράμε προς τον τομέα αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις για την κρίση. Κάνοντας το θα πρέπει να σπάσουμε την αρνητική σχέση ανάμεσα στα πιστοτικά χρέη, στα χρέη το τραπεζικά μάλλον και το δημόσιο χρέος. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει και το είχαμε πει και στο παρελθόν. Ο μηχανισμός εποπτείας των τραπεζών θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους επενδυτές και στους εμπλεκόμενους στην οικονομική δραστηριότητα γενικότερα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει επίσης και με τα συστήματα τα εθνικά εγγυήσεων ε, και αυτό θα πρέπει να γίνει στις, ε, βασιζόμενοι στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την εποπτεία των τραπεζών και τα συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων που λειτουργούν, που ισχύουν σε διάφορες χώρες. Αυτά είναι θέματα στα οποία καλείστε και εσείς να παίξετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουμε γρήγορα. Αγαπητά μέλη, Άμα πριν περάσω και σε άλλα θέματα πιο μακροπρόθεσμα, ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω τώρα με το λεγόμενο διπλό πακέτο. Εδώ πρόκειται για ένα βασικό πυλώνα. Είναι η απάντησή μας στην κρίση και ε, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται και αυτό να συμπεριληφθεί όπως και άλλα στοιχεία του Δημοσιονομικού Συμφώνου στην κοινοτική μέθοδο. Αυτό λοιπόν εμείς πράττουμε με το διπλό αποκαλούμενο πακέτο. Τώρα λοιπόν που οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και τα κρατημέλη έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία στοχασμού που αφορά όλα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης, ελπίζω θα μπορέσετε να συμφωνήσετε ότι το διπλό αυτό πακέτο έχει προτεραιότητα και δεν θα πρέπει να εξετάσουμε άλλα θέματα που αφορούν στην περαιτέρω βάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία της εμπάθυνσης ε, της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής ε, Ένωσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, καλούνται να τοποθετηθούν στην ενδιάμεση, όπως αποκαλείται, έκθεση, την έκθεση που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ε, θετική συνεισφορά του Πρόεδρου κ. Σούλτ. Πάμε στα επόμενα βήματα. Νομίζω σα έχω ήδη τον προηγούμενο μήνα ενημερώσει ότι το σχέδιό σα ε, πράγματι το καταθέσατε έγκαιρα πριν από το Δεκέμβρη. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο θα αναφερθούμε σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εμβάθυνση τη Νομισματική Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, επιτρέψτε μου να πω και λίγα λόγια που αφορούν στη δημοσιονομική επάρκεια της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης. Όπως ήδη είπα στην κατάσταση της Ένωσης όταν μίλησα εδώ, για να καταφύγουμε στην έσχατη λύση πρέπει να έχουμε ε, πλήρη και αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση, να έχουμε και μια αποτελεσματική δημοσιονομική ικανότητα της Ένωσης αυτής. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή των βασικών οικονομικών πολιτικών, κυρίως στην Ευρωζώνη, αυτό ως ένα αποτελεσματικό μέσο για να αποτρέψουμε ανισορροπίες. Ενώ πάρα πολλά γίνονται εδώ, παραδείγματο χάρη με το αποκαλούμενο εξα, εξαπλό πακέτο, περαιτέρω βήματα είναι καθοριστικά για να συνδυάσουμε συγκεκριμένες συνθήκες με συγκεκριμένα κίνητρα και για να μπορέσουμε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να γίνει βιώσιμη. Εδώ λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχουν συμβατικές ρυθμίσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αυτές θεωρούν ότι θα πρέπει να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις των κρατών των μελών, βεβαίω με συγκεκριμένη υποστήριξη για την επίτευξή του. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αποφάσει που θα ληφθούν για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ελπίζουμε θα μπορέσουμε να ε, συνομολογήσουμε τι επόμενε εβδομάδε. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σα σε όλα αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τι απόψει και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε βήμα, γιατί σχεδιάζουμε ένα νέο σύστημα όπου περισσότερε αποφάσει αποφάσεις θα λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη λογοδοσία. Η λογοδοσία να υπάρχει στο επίπεδο που λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές που θα διατρέξουν τις συζητήσεις μας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και παράλληλα οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι μεγαλύτερη δημοκρατία σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και όχι μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ήδη πολύπλοκο είναι το σύστημα λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμοί, διαδικασίε. Αυτά όμω καθιστούν την Ευρώπη λιγότερο ευανάγνωστη θα έλεγα, ε, με λιγότερη διαφάνεια. Τη στιγμή όμως που οι πολίτε και τα κράτη-μέλη πρέπει να έρθουν πιο κοντά. Και υπάρχουν ορισμένε βασικέ αρχέ των μεταρρυθμίσεων. Καταρχήν, οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε το κείμενο πλαίσιο, το νομικό, που βασίζεται στι κοινοτικέ συνθήκε. Οφείλουμε να στηρίξουμε την εμβάθυνση τη νομισματική ένωση, αυτό ω βάση για να ενισχύσουμε το ευρώ. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σύγκληση ανάμεσα στα υπάρχοντα, τα νυν και τα μελλοντικά μέλη τη ε, ευρωζώνη. Η αποφάσεις ε, ε, λαμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 27 μέλη, κυρίως ε, και σύντομα 28 και αυτό αφορά την ακαιρεότητα της κοινή αγοράς. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας παρουσίασα τα καθήκοντά μας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το διπλό πακέτο και η τραπεζική εποπτεία είναι δύο καθήκοντα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Και αναφέρομαι κυρίως στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρώ οι κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες μιλούν διαρκώς για τις επενδύσεις για να προαχθεί η ανάπτυξη και οι θέσεις απασχόλησης θα συμβάλλουν οι κυβερνήσεις αυτές έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πάλι λοιπόν αυτό θα είναι λιδία λίθος για το κατά πόσον υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Κατά τη διάρκεια των ε, συναντήσεων κορυφή, είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε και ένα μήνυμα προ την Ελλάδα ε, στο πλαίσιο τη Ευρωζώνη. Τα συμπεράσματά μα και χαιρετίζω τα συμπεράσματα αυτή τη συνάντηση, όπου είπα και παραθέτω. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα προβεί σε δημοσιονομικέ μεταρρυθμίσει και την ενισχύουμε στι προσπάθειά τη να εφαρμόσει ταχύτατα το πρόγραμμά τη. Είναι απαραίτητο έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Οι προποθέσει αυτέ θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να επανέλθει στην ανάκαμψη και θα διασφαλίσουν το μέλλον τη στην Ευρωζώνη. Τέλο τη παράθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε την προτιμία τη και τη δέσμευσή τη να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Τέλο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, τοποθετήθηκε στην εξωτερική διάστηση των πράξεών σε συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων με την Κίνα, όπω επίση και το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ατζέντα προληπτική, α πούμε, σχετικά με το εμπόριο. Εμεί ενδιαφερόμαστε για την παγκοσμιοποίηση, αλλά το να είμαστε ανοιχτοί είναι σημαντική προπόθεση για να αντιμετωπίσει κανεί την ανάπτυξη και δεν πρέπει να χάσουμε τι ευκαιρίε για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι σημαντικό σε μια εποχή όπου πολλοί πολίτες αμφιβάλλουν για τη δυνατότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, είναι σημαντικό το ότι η διεθνής κοινότητα με το ε, βραβείο Νομπέλ μας έστειλε ένα σαφέ μήνυμα ότι επιθυμούν μια ισχυρότερη Ευρώπη. Είναι λοιπόν τιμή αυτή η αναγνώριση στον δρόμο μας ε, για την πρόοδο σε αυτή την Ήπειρο που ε, εδώ και 60 χρόνια έχει φέρει και έχει επιτύχει τόσα πολλά. Είναι όμως επίσης ευθύνη ευθύνη μας και πρόκληση να επιδείξουμε καθημερινά κουράγιο στην καθημερινότητα, να κάνουμε τα σωστά πράγματα, να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Προχωρώντας λοιπόν στην εμβάθυνση της ε, νομισματικής ένωσης, βαδίζοντας προς μια πολιτική ένωση, ας διασφαλίσουμε από κοινού ότι το βραβείο αυτό του 12 δεν αφορά τις απόψεις του παρελθόντος, αλλά τις προοπτικές του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παρόσο. Ακολουθούν οι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ξεκινούμε με τον κύριο Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είμαι εκφύσεω αισιόδοξο άνθρωπο, αλλά η αισιοδοξία μου είναι και ρεαλιστική ταυτόχρονα. Στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και σε συγκεκριμένα επιτεύγματα και στην εμπειρία της τελευταίας εξεκονταετίας που τελικά είναι μια αρχή μόνο. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την αναγνώριση αυτής της κοινή μας προσπάθειας τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι και μια ενθάρρυνση όμως να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, να πάμε πιο μακριά. Πιστεύω στην Ευρώπη, πιστεύω στην κοινοτική μέθοδο στην υπεραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στις κοινέ της πολιτικέ. Πιστεύω όμως ταυτόχρονα και στην, ε, σε ευρωπαϊκές επενδύσεις στον προϋπολογισμό μας που κάθε χρόνο αφιερώνει ε, εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ευρώ στις οικονομίες, αλλά αυτό είναι λίγο. Χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξες πολιτικές. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα μας επαναφέρουν στο δρόμο της ε, οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Και για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και ένα φιλόδοξο κοινοτικό προϋπολογισμό. Και αυτό το έχει καταδείξει και η συζήτηση. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην ευθύνη όλων. Θα πρέπει όλοι να επομιστούμε ε, τις ευθύνες μας και να προβλέψουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που θα είναι φάμιλο των φιλοδοξιών μας αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αξιόπιστοι προς τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περίεσμένης εβδομάδα ε, έκανε ένα επιπλέον βήμα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής Ένωσης. Γιατί η κρίση μας είναι οικονομική. Λάθος μας όμως ήταν που δεν σεβαστήκαμε τις υποχρεώσεις μας, τις δεσμεύσεις μας και τους κανόνες που είχαμε ήδη θεσπίσει. Τους τελευταίους μήνες επομιστήκαμε τις ευθύνες μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό προβλέψαμε τους απαραίτητους μηχανισμούς. Το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση που επιβάλλει διατάξεις που θα πρέπει όμως να εφαρμοστούν. Το ίδιο ισχύει και για το διπλό πακέτο, το 2-pack που εξετάζουμε σήμερα ε, τις διάφορες του πτυχές και πιστεύω ότι θα έρθει σε αίσιο πέρας. Ένα από τα διδάγματα της κρίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι δεν μπορούμε να ε, αποκλείουμε ορισμένους τομείς από την κοινή νομοθεσία, τον τραπεζικό τομέα για παράδειγμα. Η ομάδα μου ε, είναι ιδιαίτερα προσεκτική στα θέματα αυτά. Στηρίζουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου για τη σύσταση μιας ενιαίας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν τεράστιες αλληλεπιδράσεις. Η παραμικρή αποτυχία, ε, το ελάττωμα ή το λάθος μιας μικρής τράπεζας έχει αντίκτυπο σε όλο το σύστημα. Και αν μερικές τράπεζες θεωρούνται υπερβολικά μεγάλες για να χρεοκοπήσουν, καμία τράπεζα δεν είναι υπερβολικά μικρή για να ε, εκφεύγει τη εποπτική αρχής. Πιστεύω ότι και οι επιχειρήσεις μας και οι τράπεζες μας χρειάζεται να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και το ΕΛΚ έχει αναλάβει τη δέσμευση ώστε να εξέλθουμε από την κρίση αυτή. Να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι η λύση. Εδώ και μία εικοσαετία η ενιαία αγορά εστέφθη με επιτυχία. Αλλά για να είναι βιώσιμη αυτή η επιτυχία και η φόρα θα πρέπει να την ολοκληρώσουμε, να διεκπαιρεώσουμε το έργο μα, να υποχρεώσουμε του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων να γεμίσουν τα κενά τη ενιαία αγορα Για παράδειγμα, η θέσπιση της ενιαίας αγοράς ε, στον ψηφιακό τομέα. Αν την αμελήσουμε θα χάνουμε κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε κύκλο εργασιών, σε τζίρο. Η Ευρώπη είναι ένα σταυροδρόμι και φυσικά πολλοί θέλουν ε, να την ε, περιορίσουν σε ένα χώρο ελεύθερων συναλλαγών, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης από τους ιδρυτές πατέρες, το ευρωπαϊκό σχέδιο έχει γίνει συνώνυμο ειρήνης και ευημερία και μάλιστα έχει επιβραβευθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και εδώ και μία εξεκονταετία είμαστε υπόδειγμα, παράδειγμα προς στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς, την αλληλεγγύη και να συνεχίσουμε να προσπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως ε, τις αξίες αλλά και πέραν τούτου, αγαπητέ πρόεδρε του Συμβουλίου, θα ήθελα και το έχω επαναλάβει πολλά και στην αίθουσα αυτή, εν μέσω κρίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις και φυσικά όταν λαμβάνουμε αποφάσεις βγαίνουν και κάποια λάθη. Το χειρότερο όμως σε μια περίοδο κρίσης είναι η υπερβολική αναμονή γιατί όσο περισσότερο περιμένουμε τόσο χάνουμε δισεκατομμύρια που επιβαρύνουν τους πολίτες μας. Είναι μια έκκληση προς εσάς να έχουμε καταλήξει συμφωνία για ένα πολύ καλό κοινοτικό προπολογισμό μέχρι το τέλο του έτου. Έτσι θα δείξουμε την καλή μα θέληση προ τον κόσμο αλλά και προ τι αγορέ. Καλή σα τύχη, εύχομαι και καλό κουράγιο για να φτάσουμε ε, να μας έρθετε με ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλιστές, ο κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το σημείο αυτό στο οποίο ξεκίνησε ο κύριος ε, ε, Φαν για το θέμα της ισότητας των φύλων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ έχω μια ίσως διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. Εγώ απογοήτευθηκα από την θέση που κράτησε το, το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Κύριε Φαν Ρομπό, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι με υπεκφυγές να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Εμείς έχουμε αναλάβει αυτήν την δέσμευση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα της ισότητας των φύλων. Το ίδιο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει δεσμευτεί για το θέμα αυτό. Δεν θέλουμε απλώ μια περιγραφή τη κατάσταση, μια διάγνωση ότι δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε σε θέσει ε, ευθύνη. Θέλουμε να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό το οποίο έχει γίνει δεν είναι μια λύση. Έρχομαι τώρα στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανεί να χαρακτηρίσει ω αρνητικά τα συμπεράσματά του, αλλά ήταν χλιαρά, δεν οδήγησαν σε τίποτα. Το σύμφωνο σταθερότητα. Δεν χρειάζεται να συνεδριάσουμε 28 χώρε για να καταλάβουμε ότι δεν λειτουργεί το σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό που μα ενδιαφέρει να έχουμε οικονομική μεγέθυνση. Το πρόβλημα τη ανάπτυξη δεν προέρχεται από το ίδιο το σύμφωνο. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε ακόμα να συζητήσουμε σε βάθος για τα θέματα αυτά. Γιατί δεν δέχεται η Κομισιόν αυτά τα οποία έχουν φανεί και από την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα οικονομικά προβλήματα και για τους λόγους για τους οποίους καταλήγουμε σε μια ύφεση. Δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει μια πραγματική συζήτηση. Δεν είναι μόνο το σύμφωνο σταθερότητα. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική ανάπτυξη, η οποία δεν οδηγεί σε ύφεση, αλλά σε ανάπτυξη και σε απασχόληση. Αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Βλέπετε ότι η αύξηση της ανεργίας συμβαδίζει με αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της απόρριψης της Ευρώπης. Υπήρξανε αυτά τα πυροτεχνήματα της κυρίας ε, Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Αλλά αυτά δεν θα λύσουν τα σημερινά προβλήματα. Είναι απαραίτητη η Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να γίνει τώρα η Τραπεζική Ένωση, όπως είπε και ο κύριος Σολάντ. Δεν είναι τώρα μια διαφωνία Γαλλίας και Γερμανίας. Είναι μια σύγκρουση διαφορετικών απόψεων. Η μία άποψη λέει ότι τα θεσμικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θυμηθείτε την ε, συνέλευση η οποία είχε γίνει, τη συζήτηση που γίνεται τώρα για υπερεπιτρόπους, αλλά συγχρόνως, καλά είναι όλα αυτά, αλλά συγχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία πλήττουν τις χώρες μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιρλανδία, τα προβλήματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ισπανία, την ανεργία. Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουμε να οδηγήσουμε στην αθλειότητα τους Ευρωπαίους με υπερβολική λιτότητα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τις ε, τράπεζες, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των ε, τραπεζών αλλά οι τακτικοί καθυστέρηση που ακολουθείται από την Κομισιόν δεν μα εξυπηρετούν. Να υπάρξουν διαβουλεύσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ταχείε λύσει, γιατί αλλιώ η κρίση θα γίνει πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο δυνατή στην ε, Ιρλανδία και στην Ισπανία και σε άλλε χώρε. Και πάλι θέλω να σταθώ στο κοινωνικό θέμα. Μιλήσατε για αυτό τον πέμπτο πυλώνα, κύριε Φαν Ρομπάι, για τα κοινωνικά θέματα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα κοινωνικά θέματα να τα αντιμετωπίσουμε μονάχα επιδερμικά. Κύριε Μπαρόσο, κύριε Φον Ρομπάι, λέτε βλέπουμε την κοινωνική αθλειότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Μα δεν φτάνει να διαπιστώσετε αυτό το οποίο γίνεται. Πρέπει να κάνετε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Χρειάζεται αγώνα για μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι το απαραίτητο. Εμείς χαρήκαμε για το βραβείο Νόμπελ που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που μας δίνει μεγάλη χαρά και ε, υπερηφάνεια. Αλλά δεν πήραμε, δεν έχουμε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ σε ό,τι αφορά την κοινωνική ειρήνη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακόμα παραμένει να το πραγματοποιήσουμε. Και πολλά από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε την, οδηγούν την Ευρώπη στην αντίθετη κατεύθυνση. Και τέλος για τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Κάμερον μιλάει για ένα βέτο για τον προϋπολογισμό. Αν όμως ακολουθήσει ο κύριος Κάμερον μια τέτοια ε, αντιμετώπιση, θα παραμείνουμε στα όρια του προϋπολογισμού του 2012. Αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, εντάξει, κάποιες χώρες μπορεί να μην ενδιαφέρονται για την Ευρώπη πια. Αλλά εάν ο κ. Κάμερον δεν θέλει να παρακολουθήσει τις άλλες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό του 2012 σαν βάση για, την, για το μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί όμω να είναι αυτή η κατάσταση. Ο κ. Κάμερον να θέλει να αποσύρεται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη, αλλά θέλει να έχει λόγο για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν θέλουν να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α το κάνουν αλλά α μην προσπαθούν να επηρεάζουν την άποψη που διαμορφώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν θέλουν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση αποφάσεων στην Ευρώπη, θα πρέπει να συμμετέχουν στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο κ. Κάμερον. Για τους φιλελεύθερους, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την απόφαση για την Τραπεζική Ένωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νόμιζα όμως ότι ήδη από τον Ιούνιο είχε ληφθεί η σχετική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει. Καλύτερα να αποφασίζει δύο φορές το ίδιο πράγμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρά να μην αποφασίζει τίποτα. Χαίρομαι πάντως που το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, τελικά συμφωνεί και με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι το σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις τράπεζες. Και ήταν ε, παράλογη η ιδέα να εποπτεύει μόνο ορισμένες τράπεζες. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το χρονοδιάγραμμα που επισήμανε και ο κύριος Φόμποντα. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο και θετικό, γιατί το χρονοδιάγραμμα τελικά με τι συνδέεται. Με το προεκλογικό πρόγραμμα της Γερμανίας ή το πρόγραμμα των ε, γερμανικών εκλογών. Θα πρέπει να περιμένουμε εννέα μήνες πριν αρχίσουμε να εφαρμόζουμε κάτι που ήδη ε, θα έχουμε εγκρίνει ε, στην νομοθεσία μέχρι τα τέλη του χρόνου. Προς τι αυτή η εννιάμινη αναμονή, για να ευθυγραμμιστούμε με, τις, με το χρονοδιάγραμμα των γερμανικών εκλογών και να περιμένουμε την έκβασή τους. Κάθε φορά έτσι θα πρέπει να περιμένουμε. Τις εκλογές στη Γερμανία ή μετά στη Γαλλία ή μετά στην Ιταλία, οπότε τι θα κάνουμε. Θα περάσουμε το χρόνο μας ε, μόνο σε αναμονή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγγραφο. Υπάρχουν μερικές ε, καλές ιδέες στο έγγραφο, κύριε Πρόεδρε και κάποιες προβληματικές. Το θέμα των ατομικών συμβάσεων, για παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μια ιδιωτική επιχείρηση που θα στηρίζεται σε μεμονωμένες συμβάσει διμερείς μεταξύ των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Θέλουμε γενικές πολιτικές και δεσμευτική νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά την κοινή ανάληψη του χρέους. Κύριε Μπαρόζο, Κάθε μήνα το ίδιο σας ρωτάω. Πού είναι η πρότασή σας για το Ταμείο Απόσβεσης του Χρέους και για την έναρξη της εφαρμογής των ευρωομολόγων, μιας αγοράς ευρωομολόγων. Μόνο έτσι θα μειωθούν τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Σλοβενίας. Έχει κάτω του 60% δημόσιο χρέος και ταυτόχρονα έχουν ένα δημοσιονομικό έλλειμμα 3%. Τι επιτόκια καταβάλει η Σλοβενία? 6%! γιατί είναι μια μικρή αγορά και κανένας δεν ενδιαφέρεται σήμερα σε αυτή την κρίση να αγοράσει εθνικά ομόλογα της Σλοβενίας. Μόνο με τα ευρωομόλογα θα λύσουμε αυτή την μάστιγα των υψηλών επιτοκίων. Και θα πρέπει να εθετήσουμε το διπλό πακέτο. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής πάντως. Αν δεν υποβληθεί πρόταση για το redemption φατοδομείο ε, απόσβεση του χρέους, δεν πρόκειται να εγκρίνουμε το διπλό πακέτο. Το ίδιο ισχύει για την πρόταση του κυρίου Σόιμπλε. Εκείνο θέλει τον υπερεπίτροπο για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Όχι, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Παρόλο που είμαι καταρχήν υπέρ τη πρόταση, αν δεν υποβληθεί πρόταση για κοινή ανάληψη του χρέου και πρόταση για το Ταμείο Εξόφληση του Χρέου, ε, ε, πρώτο βήμα και για αυτό και για τα ευρωομόλογα, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε και με τι υπόλοιπε προτάσει. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η μοναδική λύση για να θέσουμε ένα τέρμα επιτέλου σε αυτή την κρίση πέραν των υπόλοιπων μέτρων που θα χρειαστεί να λάβουμε. Και τέλο, κάτι τελείω διαφορετικό κύριε Πρόεδρε. Η Συρία. Νομίζω ότι είναι και, καινή η ώρα και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει επιτέλους δράση. Ο βραβευτής με το Νόμπελ Ειρήνη κάτι θα πρέπει επιτέλους να κάνει. Ξέρουμε τι χρειάζεται στη Συρία. Το συντομότερο δυνατόν να θεσπιστεί ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Για να μην μπορεί ο Ασάτ να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, να χρησιμοποιεί την αεροπορία του για να σκοτώνει το λαό του, για να σφαγιάζει του συμπολίτε του. Έχουμε καθημερινά ε, βομβαρδισμούς ε, στη Βηρητό, σαν τη Δρέσδη και άμαχο πληθυσμό που χάνει τη ζωή του. Ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε τα άλλα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, μαζί με την διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν αυτό το σκάνδαλο. Το λόγο λοιπόν εκ μέρους της ομάδας των έχει η κυρία Χάρμς. Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι, αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχήν όσον αφορά το θέμα ε, των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή τη θέση θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την κυρία Ρέντινγκ, η οποία νομίζω ότι με την πρότασή της για τις ποσοστώσεις έχει απόλυτο δίκιο όλες οι επίτροποι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια όλες οι γυναίκες που σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποκτήσει εξουσία οφείλουν να γνωρίζουν ότι βεβαίως αυτό ανάγεται στις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους αλλά επίσης και στο γεγονός ότι άλλες γυναίκες μπόρεσαν να περάσουν αυτό το εργαλείο που λέγεται ποσοστώσεις. Αυτό λοιπόν οφείλουν να το γνωρίζουν όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις. Ε, απευθύνομαι σε όλες τις γυναίκες ε, συναδέλφους και στην κυρία Ρέντινγκ προφανώς και κύριε Μπαρόζο. Από εσάς περιμένω να αναλάβετε μια θετική πρωτοβουλία που να αφορά στον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι οφείλετε να στηρίξετε την κυρία Ρέντινγκ. Όσον αφορά τον κύριο Μέρς, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι γίνονται προσπάθειες ε, να ε, υπονομευτεί η προσπάθεια της κυρίας Ρέντινγκ. Εμείς δεν θα το στηρίξουμε. Κύριε Φαν Ρόμπε, ίσως για σας να αρκεί το ότι το μέλλον των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινάει μετά το 2018. Εμάς όμως δεν μας αρκεί αυτή η προοπτική. Εμείς επιθυμούμε σήμερα να υπάρχει μία γυναίκα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτά που μας λέτε είναι η παρηγοριά, λόγια παρηγοριάς και τα απορρίπτουμε. Κυρίες και κύριοι, το βραβείο Ειρήνης εμφανίστηκε και επανεμφανίστηκε στη συζήτηση και είχα την εντύπωση ότι δεν άκουσα καλά. Άκουσα αυτήν την απόφαση του Βορρά της Ευρώπης και πρέπει να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μάλιστα το εξέλαβα κάτι το προσωπικό. Ε, ε, θεώρησα ως πολιτικός ότι μου κάνουν ε, ερωτική εξομολόγηση, μία δήλωση αγάπης σε αυτό το μεγαλεπίβολο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και πρέπει να σας πω ότι κατόπιν τούτου οι προσδοκίες μου απέναντι στην συνάντηση κορυφή είναι πολύ ψηλέ, ήταν πολύ ψηλές, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Μα πού έμεινε αυτή η έκκληση της Επιτροπής ε, Απονομής. Πού απέμειναν αυτές ε, οι προτάσεις ε, για μεγαλύτερες προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί νομίζω ότι αυτό οφείλει να σκεφτεί και αυτό, όφιλε να σκεφτεί κυρίως η Επιτροπή απονομή ε, του Βραβείου το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Κύριε Φαν Χομπέου, βεβαίως ε, Τώρα πλέον ε, υπάρχει περισσότερος χρόνος ε, σε θέματα τραπεζικής ένωσης και αυτή την πολυτέλεια μπορούμε να την επιτρέψουμε στον εαυτό μας γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν, παλαιότερα υπό τον κύριο Τρισέκ και τώρα υπό τον κύριο ε, Ντράγκη αγόρασε χρόνο. Η κρίση από πλήρη όξυνση πέρασε τώρα σε μια χρόνια κατάσταση. Όμως σας παρακαλώ μην σπαταλάτε το χρόνο και μην κάνετε αυτό που κάνατε και σήμερα με την ομιλία σας. Νομίζω ότι το τέλος Δεκεμβρίου δεν θα αφορά μόνο την Τραπεζική Ένωση. Δεν θα πρέπει μέχρι τότε η Τραπεζική Ένωση να έχει λάβει συγκεκριμένα, συγκεκριμένη σάρκα και οστά, αλλά αναφέρομαι και στους δύο άλλους πυλώνες που και αυτοί θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή η διασφάλιση των καταθέσεων και η δυνατότητα οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε όλα αυτά να εντάσσονται σε μια δημοκρατικά ελεγχόμενη διαδικασία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Τώρα, θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σβόποντα. Κύριε Ρομπέ, εσείς είπατε προηγουμένως ότι θα διορθωθούν τα πάντα το δέχομαι. Αλλά αυτό για μένα σημαίνει είτε διαβάζετε άλλα στατιστικά δεδομένα από αυτά που διαβάζω εγώ. Καλό θα ήταν λοιπόν να τα ανταλλάξουμε, αν ισχύει αυτό, εγώ από την Παγκόσμια Τράπεζα και από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Έχω στοιχεία που δείχνουν ότι η αμυγή αυστηρή πολιτική λιτότητας δεν μπορεί να εξηγιάνει ούτε καν τους κρατικούς προπολογισμούς. Στις ε, χώρες που πλήττονται από την κρίση αυξάνονται τα ελλείμματα και αυτό επεκτείνεται και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμφανίζεται εξάπλωση της ανεργίας κυρίως ανάμεσα στους νέους. Κατόπιν τούτου, εφόσον τα γνωρίζουμε αυτά, θεωρώ ότι το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την οικονομική ανάκαψη, καταλαβαίνετε ότι αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει η μέχρι τώρα πολιτική. Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από οικονομική ανάπτυξη και πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω ε, να δω τι θα συμβεί. Αυτά που είπαν ο κύριος Ταγιάννη και ο κύριος Ότιγκερ, εγώ τα εξέλαβα ως απειλή. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη 2020 σημαίνει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ε, στον ε, βιομηχανικό τομέα και αυτά που λέει ο κύριος Ότιγκερ και ο κύριος Ταγιάννη για μένα δεν υφίστανται. Κυρίες και κύριοι, τελειώντας θέλω να πω, ο πρόεδρος Ολάντ και η καγκελάριος Μέρκελ μετά τη συνάντηση κορυφής ετέθη το ερώτημα τελικά ποιος κέρδισε. Αν λοιπόν θέλετε μία απόδειξη για το ότι ε, τελικά ε, δεν απορριμήθηκε σωστά το Νόμπελ Ειρήνης, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τεθεί το εξής ερώτημα η πολιτική ένωση θα προχωρήσει από αυτούς τους δύο, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ. Η κυρία Μέρκελ πολύ πριν από τις εκλογές της θα πρέπει να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη και να εξηγήσει γιατί αυτή η πολιτική που ακολουθεί επιδεινώνει την κατάσταση και ο κύριος Ολάντ εμφανιστεί και αυτός και να εξηγήσει γιατί η Γαλλία πρέπει να παραχωρήσει την εθνική της κυριαρχία στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Σανκλέρ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαδικαστικό είναι αυτό το η παρέμβαση. Μπορεί ο καθένας να ξεπερνάει κατά δύο λεπτά το χρόνο παρέμβασή του. Θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Ο κύριος Κάλανεν για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποια καλά θετικά νέα από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποστήριξη της ενιαίας αγοράς για τα 27 κράτη-μέλη, πιο ελεύθερο εμπόριο, μείωση της γραφειοκρατίας και απόσυρση ορισμένων προτάσεων της Κομισιόν. Περιμένουμε να δούμε περισσότερη δράση για όλες αυτές τι πρωτοβουλίε και θέλουμε να σα υποστηρίξουμε, κύριε Μπαρόσο, για να προωθήσετε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Όταν πρόκειται όμω για το κύριο θέμα συζήτηση, για μια ακόμα φορά, για την κρίση την οικονομική, βλέπουμε ότι η διάσκεψη κορυφή δεν έχει δώσει αποτελέσματα και καρπού. Και εσεί, κύριε Φανρομπάκη ο κύριο Μπαρόσο, μιλήσατε τον Ιούνιο ενώπιον τη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για την ανάγκη να υπάρξει ισορροπία μεταξύ ε, λιτότητος και αλληλεγγύης. Είπατε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προχωρήσει αλλά βρίσκεται στον δρόμο της ανάκαμψης. Μα το καλοκαίρι είναι σαφές ότι μερικά κρατημέλη, σημαντικά κρατημέλη, είχαν δεύτερες σκέψεις και τα μικρά βήματα προς τα εμπρός τελικά έγιναν μεγάλα πηδήματα προς τα πίσω. Η μόνη σημασία αυτή τη διάσκεψη κορφή ήταν ότι είναι ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράθυρο ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τη δράση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσουν οι ηγέτε Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν και να καθισκάσουν πάλι τι αγορέ, χάθηκε αυτό το παράθυρο ευκαιρία. Και το χρονοδιάγραμμα για, το, για τις εποπτικές αρχές τα προσεκτικά λόγια, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι αυτή η διάσκεψη κορυφής ήταν μια υπαναχώρηση. Εγώ έχω μεγάλη συμπάθεια και για τι χώρε τη Μεσογείου και για τι χώρε τη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμω με αυτή την κατάσταση όπου καμία πλευρά δεν μπορεί να δεχθεί, ούτε η μία πλευρά θέλει να δώσει την κυριαρχία για τα δημοσιονομικά τη, ούτε η άλλη πλευρά θέλει να δώσει την κυριαρχία στο πορτοφόλι τη. Όπω είπε ο κύριο Ρομπάι, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά πρόοδο για τα θέματα αυτά της κρίσης πριν από τις γερμανικές εκλογές. Υπάρχει έλλειψη ηγεσία. Για να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα που ελέγχθη σήμερα. Όταν η Ευρώπη πήρε αυτό το περίφημο βραβείο Νόμπελ, αρχίσαν οι καυγάδες για το ποιος θα παραλάβει το βραβείο, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα είναι παρόν στο δείπνο των νομπελιστών. Όλα αυτά τα θέματα ενώ υπήρχαν τόσοι πολλοί οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα βραβείο Νόμπελ για τις ε, προκλήσεις που αντιμετώπισαν και που άξιζαν το βραβείο Νόμπελ. Θυμηθείτε τον Ντεγκόλ, τον Ρέιγκαν, ε, τον Κόλ, τον Ιωάννη Παύλο το δεύτερο. Όλοι εδώ πέρα σε αυτή την Ολομέλεια έχουν άτομα τα οποία μπορούν να βάλουν στον κατάλογο των ατόμων που άξιζαν να έχουν το βραβείο Νόμπελ. Είχαν ένα όμω βασικό στοιχείο από κοινού. Είχαν πολιτικό θάρρο. Το θάρρο να μπορέσουν να πάρουν πολιτικού κινδύνου, να παραμείνουν πιστοί στι απόψει του και να δεχτούν θυσίε. Και πώ αυτό έρχεται τώρα σε αντίθεση με τη σημερινή Ευρώπη, όπου οι σημαντικέ και δύσκολε αποφάσει καθυστερούν, τα χρονοδιαγράμματα τελματώνονται και χρονίζουν και οι πολιτικέ αποφάσει δεν λαμβάνονται. Το βραβείο αυτό Νόμπελ δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την κρίση, αλλά ουσιαστικά επειδή αποτυγχάνουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μορφή συγχαρητήριου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πράξη επίοικιας και ελεημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κάνει, δεν τα καταφέρνει καλά. Και αυτό ήταν σαφές και στην ανακοίνωση για το βραβείο Νόμπελ. Λοιπόν, να σταματήσουμε να συγχαίρουμε εαυτούς και αλλήλου ας προχωρήσουμε και ας προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης και να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάζονται για να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία και να ξεκινήσουμε και πάλι την πορεία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. <clears throat> για, τους, για την Ενωμένη Αριστερά έχει το λόγο η κυρία Τσίμερ. Κύριε, Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη Ρεμπέκα Χάρμς και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το γεγονός ότι εχθές το βράδυ ελήφθη η απόφαση αυτή την εβδομάδα να εκδοθεί η σύσταση να μην εκλεγεί ο κύριος Μέρς. Αυτό το βρίσκω σωστό ε, και για μένα είναι ένα μήνυμα το οποίο ελπίζω ότι θα στηρίξει και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι θα ήταν λάθος, απόλυτα λανθασμένο μήνυμα να δείξουμε ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να ε, είναι στα χέρια μόνο ανδρών. Οτιδήποτε είναι απαραίτητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προαχθεί η κοινωνική συνοχή, όλα αυτά γίνονται μόνο από άνδρες. Και πρέπει να πω, στην πλειοψηφία τους είναι και λάθο. Δεν αναφέρομαι στο σύνολο. Και όσον αφορά και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί αναφέρθηκε ότι στο τέλος εμφανίστηκαν δύο νικητές ε, στις ε, τηλεοπτικές κάμερες ε, και κανείς δεν έχασε. Ναι, ξέρετε ποιος έχασε. Έχασαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιτήθηκαν γιατί και πάλι η μόνη προσπάθεια ήταν να εξοικονομηθεί χρόνος. Δεν κατέστη δυνατόν να απαιτηθούν ταχύτατα οικονομικές αλλαγές. Και έρχομαι τώρα να μιλήσω για το σύμφωνο απασχόλησης. Δεν είναι δυνατόν στα απορίσματα ή στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναφέρεται ότι σε τελική ανάλυση Πρόκειται για τα προγράμματα προσαρμογής των κρατών στα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως όσον αφορά στην ε, χρηματοδότηση του ε, Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Δηλαδή, εσείς αμφισβητείτε το 25% ε, συμμετοχή στο μηχανισμό στήριξης και με τον τρόπο αυτό αμφισβητείτε το ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα κατά της φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάμε για 120 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Και επίσης λέτε ότι το βραβείο Ειρήνη Νόμπελ ε, το αξίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά κυρίε και κύριοι. Ποιο είναι το μήνυμα που θα έπρεπε να εκπέμψει το Συμβούλιο Κορυφής πρώτον ότι η έξοδος ε, ή η εφαρμογή της ε, λιτότητας, πολιτικής λιτότητας δεν σημαίνει αυτόματα ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εδώ και καιρό θα έπρεπε να έχει κατανοήσει ότι η πολιτική αυτή οδήγησε απλά ε, χιλιάδες ανθρώπων να διολυστήσουν περισσότερο στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν χρειαζόμαστε ε, το δημοσιονομικό σύμφωνο και δεν πρέπει να υπονοπέμβονται τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό σύμφωνο το οποίο να καλύπτει το 99% των ανθρώπων και ε, να μην ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία μόνο στο 1%. Δεν χρειαζόμαστε ε, μια βιώσιμη ανάπτυξη, μάλλον η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην ανακατανομή. Και επίσης ρίξτε και πάλι το βλέμμα σας στην Ελλάδα. Η τελευταία δόση αφορά η ομιλήτρα λέει 600 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξηγένση των προπολογισμών και 30 εκατομμύρια, λέει ομιλήτρια, προβλέπονται για τις τράπεζες. Στις, ε, στην Πορτογαλία 8 εκατομμύρια προβλέπονται για τον εθνικό προπολογισμό. Αυτά που είπατε δεν είναι ισορροπημένα. Αυτά λοιπόν πρέπει να ελέγξουμε. Αυτά διεκδικούμε. Και το χρονικό διάστημα εφαρμογής ε, της ε, Τραπεζικής Ένωσης, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Μην ξεχνάτε ότι εδώ εσείς μιλάτε για εθνικές τράπεζες δεν μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου τα κράτη θα μπορούν να καταφύγουν ως έσχατη λύση ε, ούτε αναφέρεστε στον ε, ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να τα διορθώσετε όλα αυτά και τότε αν θέλετε να ξαναμιλήσουμε για τα κατά πόσον άξιζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει το ε, βραβείο Νόμπελ. Ο κύριος Φαράτς έχει το λόγο. Κύριε Φαν όταν εμφανίσετε εδώ για πρώτη φορά σε μία κάπως ε, εντυπωσιακή ομιλία σας είπα ότι ήσασταν ο δολοφόνος της δημοκρατίας των εθνικών κρατών. Συνεχίζετε τον δρόμο σας, θα σας έλεγα ότι τώρα τα κάνετε ακόμα χειρότερα τα πράγματα από ό,τι στην αρχή. Νόμιζα ότι στην αρχή μιλούσαμε για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, μια ομοσπονδιακή ένωση. Οι δηλώσει σας όμως τώρα ουσιαστικά σημαίνουν ότι θέλετε την απόλυτη υποταγή των κρατών μελών σε μη δημοκρατικές και αδιαφανείς δομές στις Βρυξέλλες. Είδα τον πανικό που είχε δημιουργηθεί όταν αρχίσαν οι διασώσει. Φοβόντουσαν πολύ ότι θα υπάρξει μια οικονομική διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί όμω είδατε αυτέ τι ενέργειε διάσωση ω την ευκαιρία σα για να αναλάβετε τον έργο. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ιρλανδία ή στην Ελλάδα. Έρχονται οι εκπρόσωποι τη Τρόικα, έρχονται ορισμένοι υπάλληλοι, περνάνε κάποιε μέρε στη χώρα, κάνουν έρευνα και μετά λένε στου εκλεγμένου πολιτικού, του πρωθυπουργού τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν και βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενθουσιασμό εδώ για να γίνει το ίδιο πράγμα με την Ισπανία. Πολλοί θέλουν η Ισπανία να δεχτεί τη διάσωση ώστε και αυτοί να υποταγούν στη νέα τάξη πραγμάτων. Και στην Ιταλία ο κ. Μόντι, ο οποίο έχει διοριστεί πρωθυπουργό, θέλει η ίδια του η χώρα να διασωθεί γιατί με τον τρόπο αυτό θα ξεπεράσει αυτό τον κίνδυνο η κοινοβουλευτική δημοκρατία να απορρίψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η επόμενη φάση είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν διασωθεί και μπορεί να μην χρειάζεται να διασωθούν, θέλετε τώρα αυτοί να υπογράψουν εγγύησει, εγγύησει για τον προπολογισμό. και θέλετε να έχετε τη δυνατότητα εσείς να διαγράψετε τους εθνικούς προπολογισμού που έχουν εγκριθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωζώνη είναι ένας πολύ σκοτεινό χώρο πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά και φοβάμαι ότι η χώρα μου που είναι παγιδευμένη εκεί θα παραμείνει εκεί για κάποιο διάστημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δόθηκε το βραβείο Νόμπελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία δεν εισέβαλε στη Γαλλία μετά από το 1945 αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε και προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο, εκτός αν όλα αυτά τα οποία λέτε είναι ότι οι Γερμανοί είναι κατά βάση κακοί άνθρωποι. Όχι, η απειλή ερχόταν από τη Ρωσία και πρέπει να ευχαριστούμε τον ΝΑΤΟ που δεν ήρθε, δεν έγινε πραγματικότητα αυτή η απειλή και τα εκατομμύρια των Αμερικανών στρατιωτών που υπηρέτησαν σε ευρωπαϊκό έδαφος για να εξυπηρετήσουν την ειρήνη. Κανείς δεν λέει τίποτα για όλα αυτά γιατί όλοι αποστρεφόμαστε την Αμερική. Αλλά έχουμε τώρα μια Ευρώπη όπου ανεβαίνουν οι νεοναζί, όπου έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις στους δρόμους και εγώ πιστεύω ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ ουσιαστικά απάδει στον οργανισμό που αποδίδει το βραβείο Νόμπελ. Εδώ έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία Βρετανών που θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αφήνει τον Ντέβιτ Κάμερον να είναι ανάμεσα σε δύο απόψεις. Προσπαθεί να δείχνει ότι τα καταφέρνει πολύ καλά στην Ευρώπη και κερδίζει ε, νίκες, αλλά χάνει και την υποστήριξη εκατομμυρίων από τους δικούς του ψηφοφόρους στη Μεγάλη Βρετανία και θα πρέπει να αποφασίσει κάποτε. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα εκ μέρου ε, των ε, μη εγγεγραμμένων η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχουμε και πάλι ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που υπόσχεται μια λύση, αλλά ελάχιστα τελικά επιτελεί. Και μάλιστα μη εκλεγμένοι ευρωκράτες και θελοτυφλούντες ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν την κρίση για περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό είναι το βαρύ τίμημα που πληρώνουμε για τα Ηνωμένα κράτη της Ευρώπης. Τίποτα δεν έχετε διδαχθεί από τα παθήματά σας και... Κύριε Παρόζο, με τους απαράτσικ σας, ε, ε, μιλάτε ότι είναι δυσανάγνωστη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, πολίτες. Είδατε τι έγινε με την κατάρρευση της ε, Ελλάδας ε, και πώς έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες στη χώρα αυτή. Φαίνεται βέβαια ότι η χώρα μου εκτό Ευρωζώνη δεν έχει επηρεαστεί. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έχετε βλέψει προ την ευημερία του ΣΥΤΗ. Ε, βέβαια, είπατε ότι δεν υπάρχει επιστροφή από την Τραπεζική Ένωση. Γιατί, ποια δυνατότητα υπάρχει για να, ε, ξαναζητήσουμε, ε, να ξανανακτήσουμε μερικέ εξουσίε που έχουμε εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποσχέθηκε ο Κάμερον. Φαίνεται ότι ήταν κενά αυτά τα λογική υποσχέση. Έχουμε πάλι ένα συντηρητικό κόμμα που βέβαια. Ε, Απ' τη μια υποτίθεται ότι ε, διαφωνεί με την Ευρώπη αλλά δεν κάνει τίποτα και σίγουρα οι περισσότεροι Βρετανοί ψηφοφόροι θέλουν δημοψήφισμα και φαίνεται ότι ε, παρόλα αυτά θα ε, ανατρέψουμε την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι κάνει ο Ντέβιτ Κάμερον για το μέλλον του κόμματο και για, το, το μέλλον της χώρας. Θα πρέπει να του στείλουμε ένα στεναρό και χειρό μήνυμα ότι οι πολίτε τη μεγάλη Βρετανία ζητούν δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κασουλίδης εκ μέρους του ΕΛ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την προσέγγιση αυτή από, την κορυφή, από βάση προς την κορυφή, σταδιακά, προοδευτικά, μέσα σε μια τετραετία, αυτή η προσπάθεια για την περιχαράκωση, αυτό το πάζλ για την περιχαράκωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οικονομική, ε, δημοσιονομική και τώρα τραπεζική ένωση, αυτό το ψηφιδωτό αρχίζει και ολοκληρώνεται. Βέβαια, οι θύνοντες μερικές φορές είναι πρόθυμοι, αποφάσεις κάπως αμφίσιμες, η εφαρμογή πολύ αργή, ενώ οι αγορές αντιδρούν με ταχύτητα που δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Βέβαια, με την Τραπεζική Ένωση ζητούμε από τους φορολογούμενους ε, ζητούμε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη διάσωση. Αυτή την εντύπωση έχουν οι πολίτε. Το θέμα είναι οι τράπεζε να μπορούν να δανείζονται απευθεία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα με διατάξει που θα θεσπιστούν και με μηχανισμού ε, εποπτεία σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Αποσυνδέοντα λοιπόν το βάρο του δημόσιου χρέου των κρατών μελών από το τραπεζικό χρέο για να μην επωφεληθούν οι τράπεζες. Βέβαια, πολλές, χώρες, πολλές τράπεζες ήδη ζητά, ε, έχουν ανάγκη από βοήθεια εξαιτία των νέων επιπέδων ανακεφαλαιοποίησης και των ε, δανείων που δεν αποπληρώνονται εξαιτία της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί και αναδρομικά, να καλύψει δηλαδή και τράπεζες που ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν, ήδη ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ευχαριστώ για τη σοσιαλιστική ομάδα, κύριος Χουάν Γκόγκ. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο Κορυφής του Οκτωβρίου αποφάσισε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή των αποφάσεων του προηγουμένου <clears throat> Ιουνίου. Αλλά η Τραπεζική Ένωση θα γίνει πραγματικότητα μόνο το 2014, θα καλύψει μόνο 6.000 τράπεζες στη ζώνη του ευρώ. Θα υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων, θα υπάρχει αρμοδιότητα για την επίλυση των τραπεζών, αλλά πάλι θα πληρώσει την ύφη ο φορολογούμενος, γιατί οι πολίτες και ιδίως οι μισθωτοί δεν είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κρίση. Οι πραγματικοί <clears throat> κακοποιοί που οδήγησαν στην κρίση είναι οι άπλιστοι χρηματιστές. Και σήμερα έχουν γίνει κατήγοροι οι οποίοι κατηγορούν τους πολίτες γιατί θέλουν κοινωνική ειρήνη η κοινωνική ειρήνη είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να εξασφαλίσουμε στην Ευρώπη. Ο κοινωνικός πυλώνας και ο δημοκρατικός πυλώνας πρέπει να είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που κάνετε οδηγεί τους πολίτες να περνούν στον ευρωσκεπτικισμό. Στην έκθεση τη ΕΝ το έχει τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική και νομισματική ένωση που να επιτύχει χωρί δημοκρατία και χωρί κοινωνικό σύμφωνο. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να παρεμβαίνει, να συζητά τις αποφάσεις της Τρόικα, να μπορεί να παρεμβαίνει στις ε, διαδικασίες διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Και η λιτότητα του προπολογισμού θα πρέπει να συνδυάζεται με την δυνατότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού να αντιμετωπίζει τα ασυμμετρικά σοκ, όπως αναφέρεται και εσείς ο ίδιο, κύριε Φων Πρέπει όμως αυτό το αντικυκλικό ταμείο να τροφοδοτηθεί με νέα κονδύλια, με μόνιμα κονδύλια και να την χάνει διαχείριση μέσω της ενωσιακής διαδικασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πολλοί από εμά συμφωνούμε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει επιτυχημένη μετάβαση προς τον φεδεραλισμό χωρίς αλληλεγγύη, χωρί κοινωνική ειρήνη, χωρί δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο πρόεδρό του στι επόμενε συζητήσει. Ευχαριστώ, για τους φιλελεύθερους <clears throat> η κυρία Ντεσσαρνές για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω προς κυρίους Μπαρόζο και Βανεροπόη ότι ακούγοντας τους ε, είναι σαν να ε, ε, διαπιστώνει ένα πρόβλημα χρονισμού δεν νομίζω ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει την κρίση. Δηλαδή δεν περιμένουμε αποφάσεις και δράσεις για αύριο, για μεθαύριο. Σήμερα τις θέλουμε και έχω κάποια παραδείγματα για την Τραπεζική Ένωση. Όλοι είμαστε υπέρ εδώ της Τραπεζικής Ένωσης. Το θέμα όμως είναι να είναι αποτελεσματική και λειτουργική αυτή η Τραπεζική Ένωση ήδη από τώρα, από αύριο και όχι μέσα σε ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο για να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε το δημόσιο χρέο και όχι να το επιβαρύνουμε. Επίση, ταυτόχρονα με την Τραπεζική Ένωση χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό αλληλεγγύη και ένα, μια ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Ευρωομόλογα, αυτό χρειαζόμαστε. Γιατί πραγματικά έχουν αφεμαχθεί οι χώρε μα ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, την οικονομική πολιτική, τι επενδύσει. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε τι απαραίτητε δημόσιε πολιτικέ. Ε, καλύτερα να προλάβουμε παρά να θεραπεύσουμε. Όχι να περιμένουμε να βρεθούμε σε ύφεση για να λάβουμε τις αποφάσεις. Θα είναι πολύ αργά σε ό,τι αφορά τη ε, ισοτιμία των θεσμικών οργάνων και την συμμετοχή των δύο φίλων, ιδιαίτερα στην ΕΚΤ. Σήμερα θα πρέπει να λάβουμε τι αποφάσει και όχι το 2018. Ποια είναι η αξιοπιστία μα όταν υπερασπίζουμε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα τη γυναίκα και ε, εθελοτυφλούμε απέναντι στις δικές μας χώρες μέλη που δεν σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών. Τι γίνεται με την δημοκρατική νομιμοποίηση. Τώρα θα πρέπει να τη θέσουμε επιτάπητος, τώρα να τη συζητήσουμε και τώρα να σημειώσουμε πρόοδο. Δαμή θα χάσουμε ε, άπαξ και διαπαντός την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σέπινγκ εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ εσάς και τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Φαν Ρομπάι για τον Νόμπελ που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν μπορώ να συγχαρώ τον κύριο Βιδάλ Κοάδα, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί στην Ισπανική τηλεόραση ζήτησε να πάει η Γουάρδια Σιβίλ στην ε, Καταλωνία και να καταπνίξει την προσπάθεια ανεξαρτησία τη Καταλωνία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι οι Καταλανοί ο κύριος Κάμερον για τη σκοτική ανεξαρτησία. Τι είπε, βεβαίως σας γίνει ένα δημοψήφισμα το 2014. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα. Όχι με στρατό ή με χωροφυλακή, αλλά με τη δημοκρατία. Για να εξηγήσει τα σχόλιά του, ο κύριος Βιδάλ Κουάδρος μας έστειλε μια επιστολή που έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Έχω εδώ αυτή την επιστολή. Διαβάζοντα αυτή την επιστολή, κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι την είχε γράψει ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Φράγκο. Λέει ότι η ανεξαρτησία της Καταλωνίας δεν είναι ούτε ειρηνική ούτε δημοκρατική. Μα τι, τι μπορεί να είναι. Τι θα κάνετε εσείς λοιπόν βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ. Εσείς κύριε Σούλτς τι θα κάνετε για το θέμα αυτό. Κύριε Σούλτς είπατε ότι ο κ. Ντάρκο εξέφρασε τι προσωπικέ του απόψει. Δεν εκφράστηκε σαν αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά έτσι παρουσιάστηκε στην Ισπανική τηλεόραση και είναι 24 ώρε την ημέρα, 7 μέρε την εβδομάδα αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μην αποφεύγετε την πραγματικότητα λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ζητήστε από τον κύριο Κουάδρας να ζητήσει συγγνώμη από το Κοινοβούλιο, να ζητήσει συγγνώμη από τους Καταλανούς και να παρετηθεί. Δεν αντιπροσωπεύει, δεν αντανακλά την ε, αξιοπρέπεια της θέσης του δεν αξίζει το ε, βραβείο Νόμπελ. Θα έλεγα ντροπή, ντροπή κύριε Βιντάλ Κουάντρας, στα Ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Σίγουρα θα μιλήσετε αργότερα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέει ο πρόεδρος τον κύριο Ραπίνο. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ασο. Χατζηγεωργίου, Έχετε ένα ερώτημα στον κύριο Έπινγκ. Ναι, ναι, μια στιγμή κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Βουλευτά, χρησιμοποίησατε το λίγο χρόνο που είχατε για να πείτε πράγματα τα οποία πηγάζουν από απόλυτη άγνοια. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας είπε ότι απλώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το οποίο είναι γραμμένο στο ισπανικό Σύνταγμα. Όλα τα άλλα που λέτε είναι προσωπικές απόψεις τις οποίες εγώ μπορώ να κατανοήσω και να σεβαστώ, αλλά τις οποίες απορρίπτω τελείως. Κυρία Πινγκ, θέλετε να απαντήσετε. Το μόνο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εγώ δεν θέλω να παρεύω στα εσωτερικά θέματα της Ισπανίας, αλλά δεν εγκρίνω μια παρατήρηση από τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου που ζητά να αποσταλεί στρατό σε μια επαρχία της Ισπανίας. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί από τους ε, εκλογείς και όχι από το στρατό. Ξέρετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Ας μιλήσουμε για δημοκρατία και ας το αποφασίσουν ήδη οι Καταλανοί και όχι οι χωροφυλακοί. Κύριος Χατζηγεωργίου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει περιγραφεί εδώ με μελανά χρώματα η κατάσταση. Και έχει περιγραφεί και από τον κύριο Μπαρόζο και από τον κύριο Ρομπάη το πρόβλημα όμως είναι τι κάνουμε μετά την ανάλυση. συζητάτε με βραδείς ρυθμούς και αποφασίζετε αργά ότι θα λάβετε κάποια μέτρα πολύ πιο αργά. ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν χρησιμοποιήθηκε καλύτερα η δημοκρατία εις βάρος του δήμου και των πολιτών. λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει άμεσα η δυνατότητα κατευθείαν χρηματοδότησης των τραπεζών δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι κύπροι και οι ισπανοί θα φορτωθούν το χρέο των τραπεζών. δεν γίνεται ιδιωτικό χρέο να γίνεται δημόσιο. πόσο πιο απλά να το πει κανεί. ενώ συμφωνείτε ότι αυτό πρέπει να γίνει το αφήνετε για μετά. κάνετε ό,τι κάνατε πάντα. σκέφτεστε μόνο πάνω από ερήπια. κλείνω. επιπρόσθετα η πρόταση για το 10% ίδια κεφάλαια των τραπεζών είναι μια πρόταση η οποία σπρώχνει στο να σταματήσουν οι τράπεζε να δίνουν δάνεια. Τι άλλο από παραλογισμό μπορεί να ονομαστεί αυτό. Ευχαριστώ. E κυρία όσον αφορά το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη, θα έλεγα κύριοι εσεί που θα το παραλάβετε να αποδώσετε τι πρέπουσες τιμές στον πολίτη τον Ευρωπαίο που το αξίζει πραγματικά και αυτός είναι ο μεν πολίτης του νότου ο οποίος πλέον δεν μπορεί ούτε να επιβιώσει με τις συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει και στον δε πολίτη του βορρά τον ευρωπαίο πολίτη του βορρά ο οποίος συνεχίζει σε ένα πνεύμα αλληλέγγυας ευρώπης να στηρίζει τον νότο αυτοί οι δύο πολίτες δίνουν τη μάχη και παραμένουν σταθεροί στο ευρωπαϊκό όραμα. και κύριε πρόεδρε μια και μπήκαμε σε ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε ότι δεν μειώνονται τα ποσά των διαρθρωτικών ταμείων τα οποία προορίζονται για τον νότο και τα οποία είναι κέρια για την ανάπτυξή του. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τζαφέλα. Ο κύριος Μόλτσα εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από τη συνάντηση κορυφής είχε αναφερθεί ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις, απλά θα δρομολογηθούν προγράμματα. Αλλά αυτή η δρομολόγηση κατά την άπεψή μου απλά ε, συνεχίζει τον παραλογισμό που οδήγησε στο αδιέξοδο. Αντί λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στις ε, περιοχές που πλήττονται από να επανέλθουν στον ορθό δρόμο. Ανταυτού έγινε ε, λόγος ε, για, τα, ε, για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Βεβαίως το σύστημα αυτό της τραπεζικής εποπτείας είναι σημαντικό γιατί πράγματι η κερδοσκοπία οδήγησε στο να πρέπει να διασωθούν οι τράπεζες με χρήματα των πολιτών. Όμως η τραπεζική εποπτεία δεν θα μπορέσει μόνη της να οδηγήσει στην έξοδο από την ευρωκρίση γιατί αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρξει πλήρης μεταρρύθμιση ρύθμιση της Νομισματικής Ένωσης. Αντί λοιπόν να τραβήξουμε το φρένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει περαιτέρω το συγκεντρωτισμό. Ε, γίνεται λόγος για τα ευρωομόλογα. Αυτό όμω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ε, αμοιβεοποίηση όπως αποκαλείται του χρέους. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο κύριος ε, Μαουρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. οι κύριοι Ντόλ και Μπαρόζο. Έχετε την καλοσύνη να δώσετε σημασία στον κύριο Μάουρο γιατί κάτι θέλει να σα πει. Εξάλλου ο κύριο Μάουρο είναι μέλο τη οικογένεια σα, άρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο ευγενικοί απέναντί του. Λοιπόν, ε, ζητώ συγγνώμη από τους παριστάμενους πρόεδρους αλλά κύριε πρόεδρε της Επιτροπής Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα, πράγματι. Αλλά η εντύπωση ε, την επαύριο του Συμβουλίου ήταν ότι επικράτησε η αρχή του, ε, της ε, προσπάθειας, της ατέρμονης προσπάθειας της Πινελόπης. Σας ερωτώ λοιπόν, για να μπορεί αυτός ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας που είναι οπωσδήποτε ένας καλός συμβιβασμό να είναι αποτελεσματικός τι προτείνεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να καλέσει τα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο λογική εξέλιξη γιατί σε διάφορες χώρες έχει αναφερθεί επανειλημμένα από αξιωματούχους ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Έτσι λοιπόν οι χώρες αυτές που ζητούν περισσότερο χρόνο φαίνεται ότι δεν έχουν σκεφτεί το γεγονός ότι ο χρόνος αυτός όμως ε, σημαίνει ότι αναβάλλονται αποφάσεις και για να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις με αποφασιστικότητα πρέπει να αλλάξουν στάση. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι θετικά αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει κανείς να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα να προκύψει το συντομότερο δυνατόν. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο κύριος Γκουαλτιέρη εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών. Κύριοι Πρόεδροι, το κοινό νόμισμα χρειάζεται μια πραγματική οικονομική ένωση, όχι ένα σύστημα κανονισμών και επιθαρχίες, αλλά μια ε, οικονομική διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε οικονομικούς ε, θεσμούς κοινού. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο είναι σαφές ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελεσματικές λύσεις που να μην βασίζονται στην κοινή αυτή, ε, στον κοινό τρόπο διαχείρισης και στα κοινοτικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το, η έκφραση του ευρώ και το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν οι αρχές σωστά επαναλήφθηκαν αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε σάρκα και οστά. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, δημοσιονομική αποτελεσματικότητα για να μπορεί να απορροφήσει αυτή το σοκ τη οικονομική κρίση. Πρέπει επίση να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτή η δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να εντάσσεται στον κοινοτικό προπολογισμό, να βασίζεται στους επιπρόσθετους ίδιου πόρου. Και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να είναι απλά ένα εργαλείο για να υπάρξει ε, μια δυνατότητα κοινή διαχείριση του χρέου. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι σε μεμονωμένες συμβάσεις γιατί με τον τρόπο αυτό απλά υπάρχει εκχώρηση και παραχώρηση ε, της εθνικής κυριαρχίας και θα υπάρχει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλλειμμα. Το Κοινοβούλιο προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο, να υπάρχουν γενικοί κοινοί στόχοι, δεσμευτικοί που θα οριστούν μέσα από τη συναπόφαση έτσι να έχουμε κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια αποτελεσματικά. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση έχει σχέση με ένα όραμα με πιο ε, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Μια Ευρώπη όπου η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατια βαντιζουν βαδίζουν χέρι-χέρι και γι' αυτό λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ένας πέμπτος κοινωνικός πυλώνας. Να υπάρχει μια εκχώρηση κοινωνικών αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει και ένας σαφής οδικός χάρτη. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί αυτή η γραμμή τη λιτότητα, να αλλαχθούν ταχύτατα κατά αποφάσεις έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το συντομότερο δυνατόν αυτά που μας προσφέρουν οι συνθήκες που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να είναι εκλογές για την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλέσουμε συντακτική συνέλευση έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική δημοκρατική κυβέρνηση στην Ευρώπη και για το νόμισμά της. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, θα ε, διεκδικήσει μέχρι το τέλος ε, της προνομή του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκουαλτιέρη. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Μπόλς. Ευχαριστώ. Πόσοι πραγματικά καταλαβαίνουμε τις συνέπειες της ενιαίας εποπτικής αρχής. Έχω την αίσθηση είναι ότι είναι σαν μια τραπεζική ένωση χωρίς όμως που θα είναι light, χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις και μια νομισματική ένωση που θα έχει de facto κοινή ανάληψη χρέου σε περίπτωση συστημικών κινδύνων. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες. Στο μεταξύ για να αποφευθεί η κοινή ανάληψη χρέου, η αμοιβαιοποίηση, η ανακεφαλαιώνουμε, ε, αποκλείται να κεφαλαιώσουμε τις τράπεζες της Ισπανίας ε, και δεν ισχύει ακόμη ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός της, της Σταθερότητας. Υπάρχει όμως άλλη ρησιμότητα, οπότε προς τι σπουδή. Μήπως ε, προσπαθείτε να μας χρυσώσετε το χάπι πριν καταλάβουν οι πολίτες τι γίνεται ή πριν αναλάβει κάποια άλλη δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπω αυτό το χρονοδιάγραμμα Έχουμε μια ε, ε, νομοθετική σπουδή αλλά μια εκτελεστική κολυσιεργία. Θα πρέπει να περιμένουμε μήνες μέχρι να έχουμε έμπραχτη εφαρμογή. Και πολλά ακούγονται για την, ε, ενιαία, για την Τραπεζική Ένωση, αλλά στο CRD, στο τέταρτη πρόταση, δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Θα πρέπει να ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται και μάλιστα εκ των προτέρων. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, παρουσία των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θέλουμε μόνο λόγια και καθόλου έργα. Έχουμε πολλές ε, υποσχέσεις ωραίες ε, για, για την ισότητα των δύο φύλων, αλλά δυστυχώς έχουν παντελώς αποτύχει οικουμενικά. Ο κύριος Στάσεν, η κυρία Στάσεν, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν ανοίξει το δρόμο προς την στρατηγική του 2020 και μία εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να στουρθοκαμιλήσουμε και να αγνοούμε τα βασικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κοινό νόμισμα σε μία ήπειρο με τόσες πολλές διαφορές δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση των εξουσιών στις Βρυξέλλες η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν περαιτέρω εκχώρηση εξουσιών στις Βρυξέλλες. Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν να λάβετε υπόψη αυτά τα σημάδια που σας δίνει η κοινωνία. Δεν πρέπει να αντλήσουμε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλετε περισσότερη κρίση, περισσότερη ανεργία, περισσότερη κοινωνική ε, αναταραχή. Έχει φύγει από τις ράγες το πολιτικό εγχείρημα της Ευρώπης πια. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε όλα αυτά με την νομισματική ένωση. Ο κύριος Οντή από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν σε θέμα διαδικαστικό. Και αναφέρομαι και στην συνέλευση των Προέδρων με τη δική σας εξουσία κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν υπήρξε μια συζήτηση με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να προετοιμάσετε μαζί μας τα Ευρωπαϊκά Συμβουλία και να ακούτε τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ απογοητεύτηκα πολύ λίγα, είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ανάπτυξη, για την ανταγωνιστικότητα, καμία πρόταση για ένα μεγάλο σχέδιο υποδομών και επενδύσεων και απλώς υπήρξε μια συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα της Τραπεζικής Ένωσης. Όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι αναφέρθηκαν, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Η Γαλλία με επικυβερνήσεως φυγιών είχε κάνει προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές στο Συμβούλιο του Ιουνίου με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και πού βρισκόμαστε. Η Γαλλία είχε προτείνει να υπάρξει μία μείωση των δημοσίων δαπανών, μία μεταρρύθμιση της εργασιακής αγοράς κτλ. Δεν ακολουθήθηκαν αυτές οι προτάσεις. Στον κοινωνικό τομέα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το άρθρο 55 του συνδικών που μας επιτρέπει να υπάρχει μια σύγκληση στους κατώτατους μισθούς οι πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι 8 χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιβάλλουμε τη σύγκληση των κατοτάτων μισθών. Θα πρέπει να, να ανακτήσουμε την ε, εμπιστοσύνη των αγορών και την εμπιστοσύνη των λαών. Ο κύριος Γκερέρος Σαλόμ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήταν δίκαιο να παραβλέψουμε τις ε, θετικές αποφάσεις και την πρόοδο που επιτελέστηκε στο Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως ήταν ε, μικρή η πρόοδος και σχετικά αργή. Ναι μεν να προχωρούμε αλλά όχι με τη σωστή ταχύτητα και αυτό θα μας απομακρύνει από την υλοποίηση των στόχων μας. Κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό αυτή τη φορά και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί επανέλαβε κάποιες αποφάσεις, ε, ε, ήταν αρκετά αργό σε ό,τι αφορά την λήψη κάποιων μέτρων και την ε, έμπρακτη εφαρμογή τους και κυρίως στον περιορισμό σε μια πολιτική λιτότητα ε, ε, με πολύ σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Ό,τι αφορά την επανάληψη των ελλημένων αποφάσεων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε περίπου 30 διασκέψεις κορυφής και πολύ δύσκολα τις διαφοροποιούμε. Θυμάστε τι έγινε στο Συμβούλιο Κορυφής του Μαΐου του 2010, της λιτότητας. Ε, του Ιουνίου του 2012 και τη θυμόμαστε γιατί είναι η διάσκεψη κορυφής της ανάπτυξης. Ε, αλλά δυστυχώς ε, η, πολυ... η... η διάσκεψη κορυφής της λιτότητας έχει αναπτυχθεί περαιτέρω ενώ της ανάπτυξης έχει συρρικνωθεί. Από τα συμπεράσματα βλέπουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν εμπράκτος και ταχύτητα τα μέτρα που θεσπίστηκαν σε προηγούμενες διασκέψεις κορυφής. Διαβάζουμε βέβαια τα συμπεράσματα και βλέπουμε ότι βρίθουν ε, ε, διατυπώσεις υπέρ κάποιου ή τις επόμενες εβδομάδες και βλέπουμε ότι τελικά μόνο 100 εκατομμύρια ε, προβλέφθηκαν για ένα πολιτικό πρόγραμμα, τίποτα παραπάνω. Και σε ό,τι αφορά την ισορροπία, δεν υπάρχει αρκετό κοινωνικό περιεχόμενο σε αποφάσεις του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αρκετό κοινωνικό διάλογο, δεν λαμβάνεται αυτό δεόντω υπόψη στι εργασίε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Και εκεί υπάρχει κάποιο κίνδυνο ο κίνδυνος να επομιστούν και πάλι μόνο τους τα κράτη-μέλη την επίλυση του, προβλημάτο, του προβλήματος της φτώχειας. Ενώ θα πρέπει η λύση του προβλήματος της φτώχειας να βρεθεί πανευρωπαϊκά. Μόνο έτσι θα δώσουμε νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, υπάρχει μια παλιά αρχή που πέρασε από τη νομική στην πολιτική πτυχή. Το Pacta Sunt Servanda. Θα πρέπει να τηρηθούν τα... οι αποφάσει τα, θα πρέπει, τα συμπεφωνηθέντα θα πρέπει να τηρηθούν. Ε, στην διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου ήλθαν κάποιες αποφάσεις για την κρίση. Και ε, μετά την λήψη των αποφάσεων χαλάρωσε η πίστη στις, αγοράς, αγορές και έτσι ε, προτάθηκαν κάποιες αποφάσεις ε, για να αποσυνδεθεί το δημόσιο χρέος από, το τραπεζικό, να, να ενισχυθεί το ευρώ και να εμπεδοθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και σίγουρα το Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας ε, περιέχει κάποια θετικά σημεία. Για παράδειγμα, ε, η πρόοδο προς την Τραπεζική Ένωση. Άλλο θετικό στοιχείο ήταν η συμφωνία των 27 χωρών για την ε, θέσπιση της ενιαίας εποπτική αρχή Βέβαια, θα πρέπει και συστάθηκε η θέση της εποπτικής αρχής σχετικά σύντομα. Αλλά δυστυχώ ε, έγινε και κάποιε επαναλήψεις. Δεν ε, αρκούν ή δεν, είναι, δεν επιτρέπονται κάποιες προσωπικές ερμηνείες ε, που αλλοιώνουν την εντολή προς τους υπουργού Οικονομικών. Ούτε ε, θα πρέπει να θεωρούμε συμπεφωνημένα κάποια πράγματα που δεν έχουν συζητηθεί καν. Θέλουμε έναν ενιαίο ε, εποπτικό μηχανισμό που θα καλύπτει όλες τις τράπεζες. Επίσης θέλουμε ένα κοινό μηχανισμό ε, εγγύησης των καταθέσεων και ένα μηχανισμό για την απόσβεση της κρίσης. Θέλουμε μια πραγματική τραπεζική ένωση, κύριε Πρόεδρε. Ο Μπούλμαν για τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ό,τι και αν λέμε για τη συνάντηση κορυφή, ε, σε τελική ανάλυση εδώ που μετράει ότι η Ευρώπη παραμένει σε ύφεση. Δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχει απασχόληση και κύριε Μπαρόζο, εσεί πρέπει να αναλάβετε νέε πρωτοβουλίε ε, και κατά τη διάρκεια τη θητεία σα. Και το ίδιο ισχύει και για εσά κύριε Βαν Χομπέου. Αλλιώ η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βγει από την κρίση. Ό,τι και να κάνετε με τι συναντήσει κορυφή, τίποτα δεν θα αλλάξει. Οι νέοι τη Ευρώπη είναι άνεργοι. Και κύριε Μπαρόζο, έχετε εργαλεία. Ο κύριος Αντόρ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία, να το κάνει αυτό η Κομισιόν. Γιατί λοιπόν δεν γίνονται αυτά που πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο του εξαμήνου από τώρα και στο εξής τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να μειώσουν την ανεργία των νέων κάθε χρόνο κατά ένα ποσοστό που θα προτείνει η Κομισιόν. Γιατί να μην γίνεται αυτό δεσμευτικό. Όλα τα άλλα τα λέμε δεσμευτικά εκτός από την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Εμείς λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο περιμένουμε να αναλάβετε πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι ε, πρέπει να υπάρξουν και περισσότερες αρμοδιότητες ε, που να εκχωρηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο που το θέμα είναι ποιο ρυθμίζει τι. Και οποτεδήποτε έρχεται εδώ ο κύριος Σόιμπλε, ο Οικονομικών της Γερμανίας, ακούμε να μας λέει ότι θέλει να έχει έναν ισχυρό επίτροπο. Α το κάνει αυτό ο κύριο Ρεν. Ε, ελπίζω ο κύριο Ρεν να μα ακούει τώρα που μιλάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Κύριε Ρεν, θα ήταν θαυμάσιο να αποκτήσετε περισσότερε αρμοδιότητε. Όμω η συμφωνία να είναι ξεκάθαρη. εσεί ε, τι ε, εντολές θα τι διαπραγματευτείτε εδώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τότε θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Όχι να πηγαίνετε στι πρωτεύουσε και να σα λένε τι επιθυμούν. Εδώ να διαπραγματεύεστε διαφορετικές ε, ρυθμίσεις, όχι σε διμερές επίπεδο, όχι εδώ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει όλα τα εργαλεία, όλες τις τεχνικές και οφείλουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει. Δεν χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη, δεν χρειάζεται να οικοδομήσουμε νέα κτίρια, αυτά που υπάρχουν να τα ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση. Ε, κύριε Μπούλμαν, ε, θα στείλουμε στον κύριο Ρεν τα πρακτικά της ομιλίας σας, ε, τουλάχιστον σε γραπτή μορφή να ενημερωθεί. Κύριε Μπαρόζο, έχετε την καλοσύνη να πείτε από πίσω στον τον κύριο Ρεν που κάθεται ότι θα τον ενημερώσουμε γραπτά, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται για την κουβέντα που διαδραματίζεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα στοιχεία και τα γεγονότα είναι σαφή. Το ανέφερε και η Eurostat ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά θετικά την κρίση και ακόμα και από την ε, προηγούμενη διάσκεψη κορυφής δεν προήλθε καμία απόφαση, μόνο μερικές κατευθύνσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι φορείς για την εποπτεία των τραπεζών να μπορέσουν να αναλάβουν το έργο τους επί τη βάση των συμφωνιών το ταχύτερο δυνατό και επιπλέον πρέπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει σαφέστερες αρμοδιότητες στα θέματα αυτά. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και γι' αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συνεχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι υπολοιπόμενες του επίπεδου ευθύνη μας. Και επίσης είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη τα οποία είναι τμήματα της ε, ε, Ευρωζώνης να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι η κρίση δεν γνωρίζει σύνορα και είναι απαραίτητο η διαχείριση κινδύνου να ξεπερνάει τα στενά εθνικά σύνορα. Το ευρώ μπορεί να προστατευτεί μόνο εάν έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη και κοινή δράση. Για τις χώρες που δεν είναι ακόμα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του, συγγνώμη, της ζώνης του ευρώ, είναι πραγματικά απαράδεκτο η διαδικασία εποπτείας των τραπεζών να λειτουργεί στα πλαίσια μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων. Δεν έχουμε μάθει το μάθημα μας αν κάνουμε μια τέτοια δράση. Κύριε Γιαννάκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ορθή η στροφή προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί. Χωρίς την αναπτυξιακή διάσταση, οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης θα αποτύχουν. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι σημαντικό βήμα και μπορεί πράγματι να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη ιδιαίτερα σε χώρες που βρίσκονται σε δημοσιονομική προσαρμογή. οι πολίτες της χώρας μου αλλά και άλλων χωρών που βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει σύντομα να βγουν από αυτή την κατάσταση. όσο αφορά τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας αποτελεί πράγματι στοιχείο της εμβάθυνσης της νομισματικής ένωσης και πρέπει να επιταχυνθεί η δημιουργία του. οι τράπεζες πολύ συχνά αντί να αποτελέσουν μέρο τη λύση αποτελούν μέρο του προβλήματο. κύριε πρόεδρε ακούστηκαν εδώ σχόλια για το αν υπάρχει ισοτιμία ή όχι των δύο φύλων. πρέπει να φύγουμε από τι συζητήσει και να μπούμε στην πράξη. η ευρώπη πήρε το νομπέλ όχι μόνο για όσα έκανε στα 60 χρόνια που πέρασαν αλλά για όσα οφείλει να πραγματοποιήσει στο μέλλον και μάλιστα το άμεσο ω παράγον σταθερότητα δημοκρατία ελευθερία κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Η κυρία Τάισεν για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν πολλά μέτρα για να εξέλθουμε από αυτή την πολύμορφη κρίση. Υπήρχαν μέτρα εντός της συνθήκης, εκτός της συνθήκης, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Και αυτή είναι που χρειάζεται για να αποκατασταθεί ένα πρόσφορο χρηματοπιστωτικό κλίμα και να ενισχυθεί η απασχόληση σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανάπτυξης. Η κατάσταση φυσικά είναι περίπλοκη και απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στα κρατημέλη αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Διαβάσαμε με προσοχή τον οδικό χάρτη, το φύλλο πορείας ε, ε, που προσπαθείτε να καταρτήσετε με τους άλλους πρόεδρους κύριε Βαν για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και θα πρέπει να υλοποιηθεί γιατί η κρίση δεν πρόκειται να περιμένει τις πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεσή μου ακριβώ για αυτό τον οδικό χάρτη, για αυτό το φύλλο πορεία. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να διαβάσετε την έκθεσή μου. Εμεί προσθέτουμε και ένα πέμπτο πυλώνα στους τέσσερι που προτείνετε εσεί, ένα κοινωνικό σύμφωνο, για να μην ξεχνούμε τι είναι επίση σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την τραπεζική τράπεζα, τροποποιήσαμε αισθητά τι διάφορε προτάσει ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο και να αποφύγουμε την αργοπορία. Είναι σημαντικά αυτά τα μέτρα και θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα πρέπει όλοι να υπομισθούμε τις ευθύνες μας για να μην συμβάλλουμε και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περαιτέρω κολυσιεργία. Ο κύριος Ρανζέλ. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Κύριε, Πρόεδρε, κύριε, Πρόεδρε. του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε βέβαια έχουν μια χρονική στέρηση σε σχέση με την κρίση και αναβάλουν επίσης τη λήψη τελικής απόφασης. Υπάρχει μια βραδιπορία. Παρ' όλα αυτά, όπως σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κασουλίδης, θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μια πρόταση στον πρόεδρο του Συμβουλίου για τις χώρες που ήδη βρίσκονται υπό σύστημα διάσωσης και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι' αυτό θα θέλαμε και εμείς μια αναδρομική εφαρμογή για, τις, για τα τραπεζικά χρέη και φυσικά την αποσύνδεση του τραπεζικού χρέους από το δημόσιο χρέος. Φυσικά δεν έγινε δεκτό αυτό για την αναδρομική ισχύ. Υπήρξαν όμως κάποιες δηλώσεις από υψηλούς ηθήνοντες της Γερμανίας και της Γαλλίας λέγοντας ότι θα ε, τύχει ειδική ε, μεταχείρισης η Ιρλανδία. Δηλαδή το Συμβούλιο αποφάσισε να ε, μεταχειριστεί διαφορετικά την Ιρλανδία από ό,τι την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Επίσημα δηλαδή προτείνει το Συμβούλιο διακριτική μεταχείριση υπέρ μιας χώρας. Ο κύριος Ρόιλ. Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπη είναι τα εξή. Καταρχήν ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να προβούμε σε εξοικονομήσει. Χρειαζόμαστε επιγόντω, διαρθρωτικέ αλλαγέ ε, και κίνητρα για την ανάπτυξη. Αυτά βέβαια έγιναν και είναι αλήθεια ότι ε, η πρόοδο είναι αργή, αλλά υπάρχει πρόοδο. Και μερικού προλύσαντε δεν του καταλαβαίνω, σαν να πρέπει να επανανακαλύψουμε τον τροχό. Μα ο κόσμο είναι σωστό και καλό, Κύριε Φαν Χομπέι, σα είμαι ευγνώμων που εσεί τα τάσεστε υπέρ ε, της ε, εργασίας ε, της συνέχειας, όχι κάθε εβδομάδα να υπάρχει ένα καινούριο εργαλείο, να μην πιστεύουμε κάθε εβδομάδα ότι θα προκύψει θαύμα, συστηματική εργασία. Αυτή είναι η μόνη λύση για να προχωρήσουμε και αυτό αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες μας. Αργές αλλά σταθερές. Γι' αυτό λοιπόν η... σταθερότητα είναι σημαντικότερη από τη βιασύνη πρέπει να ελέγχουμε αυτά που ήδη υπάρχουν και όχι να πετάμε νέε ιδέε στην αγορά. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με τον τρόπο που εργαζόμαστε τώρα. Και όσον αφορά την τραπεζική εποπτεία, το θέμα δεν είναι πότε θα εισαχθεί αυτή η εποπτεία. Το είπαν αυτό και οι δύο πρόεδροι προηγουμένω. Το θέμα είναι πώ θα λειτουργεί. Και εμεί ε, πριν από αρκετό ε, καιρό λάβαμε εδώ σημαντικέ αποφάσει. σω λοιπόν τώρα ήρθε η στιγμή να εργαζόμαστε πλέον συστηματικά. Το θέμα είναι αν θα λειτουργούν, πώς θα λειτουργούν και όχι πότε θα λειτουργήσουν. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συστηματική πρόοδο, αυτή τη βραδιά, βραδία αλλά σταθερή πρόοδο. Εγώ, ε, εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι ποιος θα λέει τα καλύτερα, ποιος θα κάνει τα σημαντικότερα. Έχει κλείσει λοιπόν η συζήτηση. Ερχόμαστε τώρα στην λεγόμενη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ. Έχουμε όμως μια μεγάλη παράκληση κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε τους ε, ομιλητές από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. έχουμε πέντε λεφτά μονάχα για τη διαδικασία κάστια και έχουμε μια μεγάλη σειρά από συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Και θα κρατούσε αυτό πάρα πολύ ώρα κάνω την εξή πρόταση σε εσά να αποσυρθείτε από την αίτηση αυτή και να ακούσουμε τον κύριο Μπαρόσο και το Συμβουλίο και για τους θεατές που βρίσκονται στην, στα θεωρία των επισκεπτών. Πρέπει αυτοί οι οποίοι ακούν τη συζήτηση, να μπορούν να ακούν τι λέγεται στην Ολομέλεια και όχι να καλύπτεται ο ομιλητής από τα πηγαδάκια τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Εύσα. Παρακαλώ όλους λοιπόν να καθίσουν. Εάν δεν καθίσετε στις θέσεις δεν μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι σταματάτε τις ιδιωτικές σας συζητήσεις. Παρακαλώ σταματήστε τις ιδιωτικές σας συζητήσεις και να καθίσετε στις θέσεις σας. Παρακαλώ, η αντιπροσωπεία του ΕΛΚ κυρίως. Και η πράσινη, κύριε Άλμπρεχτ, και εσείς παρακαλώ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι μεσομακροπρόθεσμα υπάρχουν καλές πιθανότητες να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά βραχυπρόθεσμα εκείνο που υπήγει είναι η υπέρβαση της κρίσης και γι' αυτό χρειαζόμαστε ταχύτητα στις αποφάσεις με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη με σεβασμό στη δημοκρατία και συνέπεια στην εφαρμογή. και γι' αυτό κύριε πρόεδρε της επιτροπής είναι σημαντικό και το χαιρετίζουμε η απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής να υποβάλει σήμερα την πρόταση για ενισχυμένη συνεργασία για τη θέσπιση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα λίγα κοινωνικά δίκαια μέτρα που μπορέσαμε να θεσπίσουμε αυτή την περίοδο συνέπεια στην εφαρμογή είναι μια αρχή που πρέπει να ισχύει και στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. το υπογραμμίσατε για την ελλάδα και σωστά αλλά για να υπάρξει συνέπεια στην εφαρμογή δεν φτάνουν οι κυβερνητικέ δεσμεύσει. πρέπει να πιστούν οι πολίτε ότι οι θυσίε του πιάνουν τόπο γιατί χωρί του πολίτε δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχία στην εφαρμογή και σε αυτό η ένωση μπορεί να βοηθήσει εάν η ίδια είναι συνεπή στι δεσμεύσει τη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι το Συμβούλιο έχει θεσπίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Αλλά οι προτεραιότητες θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τον χώρο έρευνας της Ευρώπης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διευκόνηση της κινητικότητας των ερευνητών, να υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία, να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο και εφοροπλαίσιο έρευνας, όπως λέει και η διαδικασία της ε, Λουμπλιάνας, να φτάσουμε ένα επίπεδο 3% σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ε, έρευνας. Ξέρουμε ότι είναι νευραλγική η έρευνα για την ανάπτυξη και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα αυτό προσεκτικά στους προϋπολογισμούς. Αν μειώσουμε ακόμα περισσότερο τους προϋπολογισμούς δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα καθήκοντα τα οποία είναι απαραίτητα στο χώρο της έρευνας. Λυπάμαι για το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα έπρεπε να πάει μια αντιπροσωπεία στο Ιράν και δεν θα πάει παρόλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, οι συμπολίτες μας θα χαρούν με την αναγνώριση της ανάπτυξης από το συμπέρασμα του Συμβουλίου και της σημασίας της για το εμπόριο. Το θέμα είναι τι θα κάνετε για να πείσετε τα κράτη-μέλη να άρουν τους ε, εμπορικούς φραγμούς ώστε να λειτουργήσει πραγματικά εύρυθμα η νέα αγορά όπως επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πώς ε, θα θέλουμε τα κράτη-μέλη να ανοίξουν τις αγορές υπηρεσιών για να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Κύριε Βαρόζο, ίσως θα πρέπει να αποσύρετε κάποιες προτάσεις ε, για τη μείωση, για να μειωθεί το κανονιστικό βάρος. Γιατί προτάσεις όμως μιλάτε κύριε Βαρόζο. Χαιρόμαστε για το εξωτερικό εμπόριο και τα συμπεράσματα για την ε, Ιαπωνία, την ε, Σιγκαπούρη και την Ινδία. Αλλά μην, ε, και τη Σιγκαπούρη, αλλά μην ξεχνάτε την Ινδία και φυσικά τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και τι γίνεται με το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη. Γιατί αν ε, έχει θέληση για την υλοποίηση του στόχου, θα πρέπει να προβλέψει το Συμβούλιο και μέσα για την υλοποίησή του. Ο κύριο Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα μιλάνε για ε, ενιαία τραπεζική εποπτεία. Τι γίνεται όμως με τα ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα αποτελούν τμήμα της κρίσης. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και φυσικά η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να μπαίνει σε ξένα χωράφια. Ε, είπαμε ότι θα διαβριθούν οι αρμοδιότητες της ε, με τις αρμοδιότητες της τραπεζικής εποπτείας που όμως να διαχωριστούν από τις τραπεζικές αρμοδιότητες. Δεν θα πρέπει όμως ε, αυτή η τραπεζική εποπτεία να υπάγεται και στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξης έδειξε ότι δεν λειτουργεί επαρκώ ο πολιτικό έλεγχο, η πολιτική εποπτεία, ούτε φαίνεται ότι είναι επανάκια. Δείτε τι γίνεται στην ε, Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία. Έχουμε πραγματικά δύσκολε συζητήσει για το μέλλον του ευρώ και μερικέ φορέ θα πρέπει να έχουμε το θάρρο να λάβουμε και δύσκολε αποφάσει. Η κυρία Κουρμάη Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου ένα σχόλιο ε, που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας. Ε, ακούσαμε σήμερα την πρόταση για τις ποσοστώσεις σε Διοικητικά Συμβούλια και βλέπουμε όμως για άλλη μια φορά ότι αυτό είναι απλά ευσεβής πόθη, δεν λύνεται τίποτα. Η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα δημοκρατικό και θεμελιώδες θέμα. Κατά τα άλλα, χαιρετίζω την απόφαση των 10 κρατών των μελών να εισάγουν τον φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Η δική μας η πολιτική ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει αναπτύξει δραστηριότητα επ' αυτού. Χαιρόμαστε που αυτά λαμβάνουν σάρκα και ωστά. Επίσης η Ιρλανδική Προεδρία ε, θέλει να ε, εφαρμόσει σχετικά προγράμματα. Κύριε Μπαρόζο, είπατε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μια χαμένη γενιά στην Ευρώπη. Εσείς κύριος Βαν μιλάτε για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά διαρωτώμε πώς ακριβώς προτίθεστε να εφαρμόσετε τις πολιτικές σας αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Ο κύριος Μπάφτον έχει το λόγο. Uh, thank you, uh, President It is very rare that... Πολύ σπάνια έχω να πω κάτι θετικό για την Κομισιόν και τους Επιτρόπους. Σήμερα είναι διαφορετικά μας τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα στο κανάλι Sky News ο Επίτροπος Εμπορίου Κάρελ Ντεχούχτ δήλωσε ότι το, Ευρωπαϊκό, το, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιβιώσει χωρίς την Ευρώπη. Αυτό το λέμε εμείς χρόνια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαρόσο όταν λάβει το λόγο εάν συμφωνεί με τον Επιτροπό του. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής είναι η κυρία είναι δυνατό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη την παραδοχή των σφαλμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όταν έκανε τον υπολογισμό με τους πολλαπλασιαστές και το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής λιτότητας. Και αυτό σημαίνει ότι οδήγησε στην τραγική κατάσταση του λαού της Ελλάδος, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ιταλίας και της Ισπανίας συνειδητικά και έτσι έχει αποδυναμώσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πώς η, η Κομισιόν που είναι θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών ε, συμφερόντων δεν πιέζει την Τρόικα να επανεξετάσει τα προγράμματα προσαρμογής στο φως της παραδοχής του σφάλματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των συστάσεων της κοιλίας Λαγκάρτ να δοθεί περισσότερος χρόνος και να επιτευχθούν λογικά επιτόκια για τις χώρες αυτές. Πώ μπορεί το Συμβούλιο και η Κομισιόν να συνεχίσουν να επιμένουν σε μία συνέχιση της λιτότητος ενώ όπως το είπε πολύ σωστά ο Φρανσούα Ολάντ για τις χώρες διάσωση που είναι τόσο δύσκολη η πολιτική και η οικονομική τους κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει αυτό Αλλιώ θα έχουμε σοβαρές συνέπειε για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Γκόμε. Πολύ ωραία λοιπόν λέει ο Πρόεδρος. Έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας παρακαλέσω κυρίες και κύριοι να καθίσετε. Καθίστε παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη να καθίσετε. Κυρία Γκουρμάη, αν έχει την καλοσύνη, καθίστε παρακαλώ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπαρόζο που θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την αποτίμηση αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ακούσετε στην αρχική μου ομιλία ότι παρέπεψε σε τρία Ευρωπαϊκά Συμβούλια και το έκανα εσκεμένα γιατί το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σημαντικό γιατί και επιβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις και υπήρξε και κάποια πρόοδος. Γιατί στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες για τη δέσμευση ορισμένων κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά οι λιμένες αποφάσεις προηγούμενου Συμβουλίου. Γι' αυτό και χρειάστηκε η επιβεβαίωση. Η οριστική απόφαση για τα πιο σημαντικά ζητήματα όμως θα γίνει μεταγενέστερα. Για παράδειγμα για την ΟΝΕ το Δεκέμβριο και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ευελπιστούμε να ληφθεί απόφαση το Νοέμβριο. Οπότε ο δικός μου απολογισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι σίγουρα συνιστά πρόοδο γιατί επιβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις αλλά δεν έδωσε μία πλήρη απάντηση ε, στις τρέχουσες προκλήσεις ε, είτε της Ευρωζώνης είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι ένας ε, δίκαιος απολογισμός του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βέβαια θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ασχολούμαστε με εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα. μεγάλη απόκληση αρχικά απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι είναι προ όφελο και προ το συμφέρον όλων των θεσμικών οργάνων να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο κλίμα και τι όριμε προποθέσει για λειτουργικέ αποφάσει και συνένεση. Σημειώθηκε κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Και χαίρομαι γιατί και από τη σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο φάνηκε ευρεία συνένεση ω προ τι αρχέ που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπεριλήφθηκαν και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τράπεζες, θα πρέπει να είναι ανοιχτός όσο γίνεται και να υπάρχει πλήρης συμμετοχή και μη χωρών Ευρωζώνης αν το επιθυμούν και επίσης θα έχει θεμελιώδη κεφαλαιώδη σημασία για να μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να βαθύνει την ΟΝΕ και να διανοιχθεί ο, ο δρόμος για τις αποφάσεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Χαίρομαι για τις προτάσεις ε, της έκθεσης ε, Tyson σε ό,τι αφορά την προώθηση και την επίσκεψη των ε, εργασιών για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για να τις οριστικοποιήσουμε μέχρι τα τέλη του 2012. Σίγουρα θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας για να βελτιώσουμε τις προτάσεις του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και να περάσουμε σε μια σταδιακή λειτουργική φάση από το 2013 όπως πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινώντας με συστημικές τράπεζες και φυσικά στη συνέχεια δεχομένως επεκτείνοντας σε όλε τι τράπεζε της Ευρωζώνης αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης αν το επιθυμούν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που επισημάνθηκε, αν δεν κάνω λάθος το ανέφερε και ο κύριος Μάουρ, είναι ε, κατεπήγον χαρακτήρα τη κατάσταση. Ε, η, αίσθηση της εκτάκτου ανάγκης. Νομίζω ότι το επισήμανα και εγώ αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι και δίκαιοι τον απολογισμό μας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν όλα τα κρατη την ίδια αίσθηση της έκτακτης ανάγκης. Ίσως εξαιτία της διαφοράς της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής τους κατάστασης. Πάντως νομίζω ότι είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της αντίδρασής μας να έχουμε κάνει σωστή προεργασία γιατί ορισμένα θέματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα και δύσκολα και από τεχνική και από πολιτική άποψη, αλλά οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν όσο πιο επιγόντως γίνεται. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά το κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη και πώς ε, μπορούμε με αυτό να συμπληρώσουμε τις ε, άλλες αποφάσεις λαμβάνοντας ε, δεόντως υπόψη την κοινωνική διάσταση. Τα στοιχεία του κοινωνικού συμφώνου ήδη σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Μην ξεχνάτε ότι η στρατηγική αυτή μιλάει για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού. Και μάλιστα στο δεύτερο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών αποτέλεσε ένα απόσπαστο τμήμα της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής. Κάτι που φυσικά προπέθεσε και μια εξασφάλιση ε, τη σωστή ε, λήψη υπόψη των εργασιακών ε, θεμάτων και των κοινωνικών θεμάτων στο νέο πλαίσιο. Η ολοκλήρωση αυτή και η συμπερίληψη αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη και τα κοινωνικά θέματα αποτελούν τις διόψεις του ίδιου νομίσματος μαζί με τις επενδύσεις. Πολλοί μίλησαν ότι θέλουμε ένα πραγματικό Υπουργό Οικονομικών στην Ευρώπη. Ίσως θέλουμε και ένα πραγματικό υπουργό εθνικής οικονομίας, κοινοτικής οικονομίας για να συμπληρώσουμε το έργο μας για την χρηματοπιστωτική, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Χρειαζόμαστε μια δέσμευση για ανάπτυξη, αηφόρομος ανάπτυξη, που θα συμπεριλαμβάνει και την οικονομική αλλά και την κοινωνική διάσταση. Γιατί δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κοινωνικό αποκλεισμό ή σε κοινωνική διχόνοια μετά τις προτάσεις αυτές. Είναι σημαντικά τα κοινωνικά θέματα και οι αξίε κοινωνική ε, δικαιοσύνη, αλληλεγγύης και ίσων ευκαιριών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο τη ευρωπαϊκή ε, οικοδόμηση και να θεωρηθούν ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μελλοντική μας οικονομική ευημερία, για την ευμάρεια των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και για την ευρωπαϊκή συνοχή. Και φυσικά θα πρέπει να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και του αναπτυξιακού μας θεματολογίου. Θα υποβάλουμε σε αρχές του 2013 ένα πακέτο για την ανάπτυξη και τη συνοχή με κοινωνικά στοιχεία που, που προέρχονται και από το δικό σας κοινωνικό σύμφωνο. Σας διαβεβαιώ ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο για να περιλάβουμε και την οικονομική και την κοινωνική διάσταση στις ευρύτερες προσπάθειές μας αναχέτησης ε, της σημερινής οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές ε, λύσεις και αντιδράσεις, σε ό,τι αφορά την αμοιβεοποίηση, την κοινή ανάληψη του χρέους, γνωρίζετε τη θέση μας, ε, τη δηλώσαμε και μάλιστα και στο blueprint που σας ανέφερα, στο αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις θέσεις Δεν συμφωνώ πάντως με εκείνους που λένε ότι είναι υπέρ του περιεχομένου του διπλού πακέτου, του ΤΟΥΠΑΚ, είναι υπέρ μιας μεγαλύτερης ελοκλήρωσης τη εποπτείας τη δημοσιονομική πολιτική. είναι υπέρ τη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη κοινοτικής μεθόδου και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης Άρα παρόλα αυτά δεν θα εγκρίνουν το διπλό πακέτο αν προηγουμένω δεν ληφθούν αποφάσει όπω για το Ταμείο Απόσβεση του Χρέου, για παράδειγμα. Λάθο κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν εξαρτήσετε μια πολύ σημαντική πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από την α, συμφωνία άλλων θεμάτων για τα οποία δεν έχει οριμάσει ακόμη το κλίμα, ουσιαστικά θα παραλύσετε την οικονομική πρόοδο και την, ε, την πρόοδο στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό η θερμή μου συμβολή προς τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις είναι να υποστηρίξετε οποιαδήποτε πρόταση που θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβω όσο το δυνατό περισσότερα στην κοινοτική μέθοδο και στις αρμοδιότητες των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και σίγουρα η, η απόφαση του διπλού πακέτου εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Ένα άλλο θέμα που σας ανέφερα είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά κάποιες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα να αποσαφηλίσω και αυτό το θέμα ένας από τους λόγους της σημερινής κρίσης είναι όχι εξαιτίας της Ευρωζώνης όπως ε, υπενήχθησαν μερικοί ευρωσκεπτισκιστές. Έχουμε σήμερα την κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία εξαιτία υπέρογκου ε, δημόσιου χρέους κάποιων κυβερνήσεων και έλλειψη βιωσιμότητας κάποιων τομέων και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν η Ευρώπη η αιτία του προβλήματο, δεν ήταν η Ευρώπη η ρίζα του κακού, αλλά η Ευρώπη ήταν το θύμα του προβλήματο και προσπαθεί τώρα να γίνει τμήμα τη λύση του προβλήματο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήταν η ανεύθυνη συσσόρευση δημόσιου χρέου ε, των κρατικών αρχών και μερικέ φορέ η ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων ε, ε, φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Και δεν ήταν Ευρώπη το πρόβλημα. Κύριε Φαράζ, η χώρα σα που δεν είναι μέλο της Ευρωζώνης εφαρμόζει τώρα ένα δύσκολο πακέτο λιτότητας. Και οι Βρετανοί υποφέρουν από τις συνέπειες προηγούμενων λαθών. Δεν ήταν το ευρώ που δημιούργησε το πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε και από ε, διανοητική αλλά και από πολιτική άποψη είναι ανέντιμο να χαρακτηρίζεται το ευρώ ως την αιτία του κακού. Ίσα ίσα προσπαθεί το ευρώ να γίνει λύση του, μέρος της λύσης του προβλήματος. Και χωρίς την προσπάθεια αυτή Ούτε και οι χώρες, κάποιες χώρες εκτός Ευρωζώνης δεν θα μπορούσαν ε, να είναι λειτουργικές, να κρατήσουν το κράτος ε, πρόνοιας, ε, την δημόσια εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Η Ευρώπη είναι τμήμα της λύσης και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθεροποιήσουμε την Ευρωζώνη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Τι είδους ανάπτυξη εννοώ, φυσικά αηφόρο ανάπτυξη. Όχι ανάπτυξη με υπέρογο χρέος. Ανάπτυξη με υπέρογο χρέος δεν είναι βιώσιμη ε, μια ανάπτυξη που θα τροφοδοτείται από, από ανεύθυνο ιδιωτικό δανεισμό δεν είναι αηφόρος και βιώσιμη. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και η ΕΚΤ, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπέρ μιας δημοσιονομικής εξυγίανσης. Συμφωνώ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και οι χώρες που έχουν περιθώρια να προωθήσουν την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την σε σχέση με την εσωτερική του ζήτηση μπορούν να το κάνουν. Και σε άλλες χώρες ε, θα πρέπει να γίνει μια ε, σωστή προσαρμογή των στόχων. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και συμφώνησε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Εμεί προτείναμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία παράταση κατά ένα χρόνο για να υλοποιηθούν οι στόχοι τη δημοσιονομική εξυγίαση. Ήταν δική μα πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Πρώτα για την Ισπανία και μετά για την Πορτογαλία. Η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο παράταση κατά ένα χρόνο την ε, προσπάθεια επαναφορά ε, και διόρθωση του υπερβολικού χρέου. Και με του δημοσιονομικού κανόνε μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο. Και όταν η κατάσταση είναι ε, χειρότερη από την αναμενόμενη και η μείωση, ε, γίνεται μια διαρθρωτική μείωση του χρέους, μια παράταση για τη διόρθωση του ονομαστικού χρέους μπορεί να χορηγηθεί. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν γίνεται αυτόματα. Η κατάσταση θα πρέπει να αξιολογηθεί περιπτωσιολογικά. Αυτή ήταν η θέση και της ε, κυρίας Λαγκάρτ όταν είπε όταν είναι δυνατό και εφικτό. Όπου είναι δυνατό και εφικτό αυτή ήταν η θέση της κυρίας Λαγκάρτ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε περίπτωση χωρών που είναι υποδιάσωση, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία, θα πρέπει να, ε, να αξιοποιήσουμε τις συνέπειες μιας πιθανής παράτασης ε, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Για μια παράταση του, της παράτασης αυτής μπορεί να αυξήσει το λόγο του δημόσιου χρέους και να δημιουργήσει με αυθύνουσα πορεία και να καθυστερήσει τη χώρα το, την, το χρόνο επαναφοράς αυτών των χωρών στις αγορές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις σε τελική ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσει μόνο υποβάλλει, αλλά σε τελική ανάλυση, σε τελικό βαθμό τις, προ... τις αποφάσεις τις αναλαμβάνουν οι χώρες. Είναι έτοιμες οι χώρες της Ευρωζώνης να χορηγήσουν επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Αυτό σημαίνει για τις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα διάσωσης, η δυνητική παράταση των προγραμμάτων υπόκειται στις, ε, στους περιορισμούς που προέρχονται από το υψηλό επίπεδο χρέους. Και αυτές ακριβώς είναι και οι απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το γνωρίσουμε και δεν έχουν δώσει όλη την πρέπουσα προσοχή στο θέμα αυτό. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι λένε τώρα ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη ευκαμψία σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους είναι ακριβώς οι ίδιοι οι οποίοι προτείνουν την σκληρή αναδιάρθρωση του χρέους. Κάποιοι θεωρούν ότι μερικές χώρες δεν θα έπρεπε να είναι στη ζώνη του ευρώ. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να τονίσω. Δεν συμφωνούμε με κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσουμε την ακαιρεότητα της ζώνης του ευρώ. Γιατί αν, επειδή, αν αποδεχτείτε μεγαλύτερη ευκαμψία στις δημοσιονομικές προτεραιότητες, προσαρμογές θα πρέπει να σκεφτείτε ποιε είναι οι συνέπειες σε σχέση με την σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες που είναι υποδιάσου να ξαναγυρίσουν στην αγορά, στις χρηματαγορές για να χρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο θέλω να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα λέγοντας ότι πολλά παραμένουν να γίνουν αλλά είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Αυτοσυμβούλιο ήταν ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο όπου συζητήθηκαν όλες οι δυσκολίες με ανοιχτό τρόπο. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν ενώπιόν μας και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρονική στιγμή όπου επειδή υπάρχει λιγότερη πίεση από τις αγορές η έννοια του κατεπήγοντος σε όλες τις χώρες μας δεν είναι ομοιόμορφη. Γι' αυτό περιμένω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν, ως ευρωπαϊκούς φορείς να διατηρήσουν την για διάταξή τους και να κατανοήσουν ότι χωρίς μια πλήρη και συνολική λύση για τα θέματα διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ δεν θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη <clears throat> και η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την επανάκαμψη των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και αυτό είναι ο τελικό μα στόχο, η ανάπτυξη και η απασχόληση, αλλά πρέπει να είναι μια βιώσιμη απασχόληση που βασίζεται σε βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ε, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βαν Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί από εσά έχετε λάβει το λόγο για να πείτε ότι πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε τώρα. Εγώ σας έχω δώσει μια γενική επισκόπηση, την οποία γνωρίζετε ήδη όλων αυτών τα οποία έχουμε πράξει τα δύο και τρία τελευταία χρόνια. Ακόμα και Πολλοί από εσά είπανε, έχουν γίνει πολλά, αλλά τώρα πρέπει να θέσετε σε εφαρμογή αυτά που έχετε αποφασίσει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε νέου φορεί, νέα εργαλεία, το έχετε τονίσει, μέχρι ότου καρποφορήσουν τα εργαλεία και οι φορεί που έχετε δημιουργήσει και τεθούν σε εφαρμογή. Και μα λέτε συγχρόνω πρέπει να δράσουμε, να δράσουμε τώρα. Μα αυτό κάνουμε. <clears throat> το λέω πολύ συχνά. Αυτά τα οποία έχουν γίνει πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Όλο το έργο σας για την οικονομική και νομισματική έρευνα, το έργο που κάνετε και εσείς και εμείς, πρέπει να το διαπιστώσω ότι όλα αυτά που έγιναν και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στη θαυμασία εκτέστη της κυρίας Τίσεν, είναι πράγματα τα οποία τα αναγνωρίσατε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στην Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα, αλλά έχουμε ήδη διατρέξει σημαντικό δρόμο. Αυτό το οποίο όμως έχουμε υποτιμήσει και εκεί που πρέπει όλοι να δηλώσουμε την ενοχή μας και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών είναι το γεγονός ότι έχουμε υποτιμήσει την έκταση και το βάθος και τη σοβαρότητα της κρίσης σε όσοι μέσα από τις χώρες μας η απώλεια ανταγωνιστικότητος, η έλλειψη βιωσιμότητας του χρέους ήταν τόσο μεγάλη που θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή. Δεν θα πρέπει να φανταστούμε ούτε για μία στιγμή ότι με ένα έλλειμμα 15% του ΑΕΠ σε ορισμένες χώρες με ένα ε, χρέος 160% του ΑΕΠ ότι μπορούμε να ξεφύγουμε την ε, λιτότητα, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις ανάγκες διορθωτικών πολιτικών και πολιτικής πειθαρχία του προϋπολογισμού. Αυτή η πολιτική δεν επιβάλλεται καταρχήν από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ίδια τα γεγονότα. Είναι σαφές ότι είναι το αποτέλεσμα μιας κακής οικονομικής διακυβέρνησης και της ολιγορίας χωρών οι οποίες δεν έδρασαν εγκαίρως και ούτε συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαίρως έχει αναλάβει τις ευθύνες της. Οι πολιτικές λοιπόν λιτότητας δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται εκ των άνω προς τα κάτω. Είναι μια πολιτική η οποία ήταν αδύρυτη, αναπόφευκτη λόγω των γεγονότων. Και πράγματι όλοι μας έχουμε υποτιμήσει την έκταση και την σοβαρότητα της κρίσης. Κάναμε πολλά πράγματα παρόλα αυτά. Κάναμε πολλά πράγματα τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο οι τέσσερις πρόεδροι των θεσμικών οργάνων εργάζονται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υπάρχει <clears throat> ένα νέο πλέγμα πρωτοβουλειών, ένας από τους βασικούς πυλώνες στην διαδικασία αυτή είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Στην αρχή της κρίσης δημιουργήσαμε τρεις-τέσσερις φορείς, αλλά ήταν κυρίως σε επίπεδο συντονισμού. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία θεσμών οι οποίοι είναι πολύ πιο ευρωπαϊκοί, πολύ πιο κοινοί για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με την ενιαία τραπεζική εποπτεία η οποία θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο και μια τομή στα θέματα αυτά. Πρέπει πράγματι να εργαστούμε σοβαρά. Πήραμε μια σειρά από, από, αποφάσεις τον Ιούνιο και η Κομισιόν στη συνέχεια το Σεπτέμβριο έθεσε τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις της και το Συμβούλιο του Οκτωβρίου οδήγησε σε σημαντικές κατευθύνσεις για να εργαστούν οι αρμόδιοι υπουργοί και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις ευθύνες του για την εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης και είναι ήδη πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το ε, έργο για να είμαστε έτοιμοι στο τέλος του χρόνου. Όταν είναι έτοιμο το νομοθετικό πλαίσιο, τότε θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στο λειτουργικό έργο για την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των δομών ε, ενιαίας εποπτείας για τον τραπεζικό τομέα και θα χρειαστούν και κάποιοι μήνες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτή η εποπτεία. Βήμα-βήμα, αλλά με έναν τρόπο σοβαρό και σταθερό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να δημιουργηθεί αυτός ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, ο οποίος θα έχει ευρωπαϊκό και ενωσιακό χαρακτήρα. Λέτε να δράσουμε, πράγματι δράτουμε, αλλά με τρόπο ο οποίος είναι σοβαρός και υπεύθυνο και ο οποίος εξασφαλίζει την ποιότητα των ενεργειών μας. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, οφείλεται στην ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί. Τονίζω λοιπόν από τη δική μου πλευρά ότι έχουμε πράξει πολλά και εξακολουθούμε να πράττουμε πολλά τα οποία σε σχέση με το παρελθόν είναι σχεδόν επαναστατικά όταν μιλάμε για τους νέους φορείς και θεσμούς που θα δημιουργήσουμε. Είμαστε στο τέλος του δρόμου, όχι ακόμα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την προοπτική του τέλους του έτους, του Δεκεμβρίου. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, το έργο αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμαστε. Γιατί τώρα μετά από όλα αυτά που έχουμε κάνει και ελπίζουμε ότι και το δίπτυχο, το TUPAC θα μπορέσει να ε, εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό με επίσης όλα αυτά τα οποία έχουμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και το Σύμφωνο Ανάπτυξης με όλα αυτά που έχουν γίνει για το μηχανισμό οικονομικής αρρωγής. Μετά από όλες αυτές λοιπόν τις προσπάθειες τους διάφορους αυτούς τομείς φτάνουμε στον βασικό πυρήνα της κυριαρχικότητος και της αλληλεγγύης. Το επόμενο στάδιο θα είναι ένα ποιοτικό άλμα και το οποίο θα το επιτύχουμε σταδιακά και σίγουρα η συζήτηση που θα χρειαστεί θα είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα είναι εύκολη ούτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε σε άλλους χώρους. Όσο περισσότερα επιτυγχάνουμε, όλο πιο δύσκολο θα είναι να προχωρήσουμε περισσότερο χωρίς να θίξουμε ορισμένα ταμπού τα οποία είναι πολύ κοντά στην έννοια και της κυριαρχικότητας και της έννοιας της αλληλεγγύης και σας προειδοποιώ μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου θα έχουμε να φέρουμε σε πέρα ένα πολύ δύσκολο έργο και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα θίξουν πολλά από αυτά τα ταμπού. Μιλήσαμε για ένα πέμπτο πυλώνα, ένα πέμπτο ακρογωνιαίο λίθο. Αλλά η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε πράξει αυτό στη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Ο κύριος Μπαρόσο και εγώ αγωνιστήκαμε για να υπάρξει αυτός ο πέμπτος στόχος του αγώνα κατά της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν απόλυτα εναντίον μιας τέτοιας ρήτρας. Και παρόλα αυτά το ενσωματώσαμε στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και απασχόλησης. Τι είναι πέρα από μια κοινωνική διάσταση, τι πιο κοινωνικό είναι. Μπορούμε να πράξουμε πέρα από το να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης σε δύσκολες συνθήκες. Η κοινωνική διάσταση λοιπόν βρίσκεται παντού, σε όλες τις ενεργειές μας. Όταν πρότεινα αυτά τα τέσσερα βασικά συστατικά της πολιτικής μας, αυτά είναι τα στοιχεία που είναι παραδοσιακά παρόντα σε όλες τις οικονομικές και νομισματικές ενώσεις όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση δεν έχουν αμφισβητήσει αυτά τα τέσσερα στοιχεία αλλά συγχρόνως εργαζόμαστε και για την κοινωνική διάσταση στο εσωτερικό αυτών των τεσσάρων βασικών δομικών λήθων. Μα είναι τα κράτη-μέλη για τα οποία είναι η πιο σημαντική κοινωνική πολιτική. Πρέπει τα ίδια τα κράτη-μέλη να πάρουν τι αποφάσεις για την εξυγίανση των προπολογισμών τους. Εγώ υπήρξα Υπουργό Οικονομικών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κάθε μέτρο θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τον κοινωνικό του αντίκτυπο και θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία, αυτοί να επομίσονται και το μεγαλύτερο βάρος. αυτό είναι ο γενικό κανόνα. Πολλέ φορέ είναι δύσκολη όμω η εφαρμογή του. Αλλά η κοινωνική διάσταση βρίσκεται σε όλε τι ενέργειες και στην ευρωπαϊκή πολιτική και στην πολιτική των κρατών μελών. Λένε ορισμένοι, πρέπει τώρα να δράσουμε για την οικονομική μεγέθυνση. Μα αγαπητοί μου συνάδελφοι, η νομισματική πολιτική δεν μπορώ εγώ να κρίνω αυτή τη στιγμή, αλλά η νομισματική πολιτική με επιτόκια τα οποία είναι σχεδόν μηδενικά ή αρνητικά δεν είναι μια περιοριστική πολιτική. Με μια κεντρική τράπεζα η οποία δίνει ρευστότητα αφιδός ένα τρισεκατομμύριο ευρώ συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Όλα αυτά δεν αποτελούν μια περιοριστική, μια σφιχτή νομισματική πολιτική. Η πολιτική τώρα του προϋπολογισμού. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ελλείμματα, θα περάσουμε στο deficit spending, θα έχουμε ελλείμματα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όχι. Προσπαθούμε να απαλύνουμε τις προϋποθέσεις και για την Ισπανία και για την Πορτογαλία και για τις άλλες χώρες. Αν δεν συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή εξυγίανσης των προϋπολογισμών, οι αγορέ δυστυχώς θα τιμωρήσουν τις χώρες αυτές άμεσα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε κερδίσει με το να απαλύνουμε τους περιορισμούς θα τα χάσουν αμέσω οι χώρες αυτές με επιτόκια που θα ανέλθουν. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. Το πιο σημαντικό βραχυπρόθεσμα είναι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη για τη ζώνη του ευρώ. Και συγγνώμη που σας λέω ορισμένα στοιχεία οικονομικά, αλλά όταν λέγεται κάτι πολιτικό πολλές φορές θεωρείται ότι δεν είναι καν πολιτικά ορθό να το λέει κανείς, να το αναφέρει. Όταν βλέπω όμως την ψαλίδα μεταξύ των επιτοκίων για τα δεκαετή ομόλογα στις περισσότερες χώρες μας και τα γερμανικά ομόλογα, όταν βλέπω την τωρινή κατάσταση και τη συγκρίνω με την κατάσταση που είχε φτάσει στο απροχώρητο τους τελευταίους 12 μήνες, εγώ βλέπω να υπάρχει μία μείωση κατά 239 μονάδες βάσης στην Ιταλία, 249 στην Ισπανία, στην ε, Πορτογαλία σχεδόν 800 μονάδες βάσης, 900 στην Ιλλανδία και 270 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το να πει κανεί λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, αυτό δεν είναι σοβαρό. Ελπίζω θα είναι μόνιμε αυτέ οι σημειώσει και σίγουρα πρέπει να δεχτούμε το δίδαγμα του παρελθόντο ότι κάναμε λάθο στο παρελθόν και δεν είμαι ο μόνο ο οποίο κάνω λάθη. Τουλάχιστον εγώ το αποδέχομαι. Ορισμένοι από εσά δεν το αποδέχεστε πάντα. Αλλά είναι αυτό ένα σαφέ μήνυμα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε περισσότερη πρόοδο για την ανάκτηση τη εμπιστοσύνη. Και αν μπορούμε να να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση τότε και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα κερδίσουν από αυτή την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια αυτής της ασθενούς ακόμα ανάπτυξης στο τέλος του 2012 και στην αρχή του 2013. Το να επαναφέρουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να πράξουμε για να έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη το ταχύτερο. Αυτά λοιπόν. Αυτό είναι και το έργο το οποίο αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια φιλοσοφία σταδιακής προόδου με μικρά βήματα. Αυτό που κάνουμε όμως κάθε φορά είναι να συγκρίνουμε αυτά που γίνονται με αυτά που έγιναν στο παρελθόν και έχουμε πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα στο παρελθόν. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, ελπίζω μαζί σας τον Νοέμβριο θα μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να έχουμε όμως μια συμφωνία χρειάζεται κάτι το οποίο είναι απαράγραπτο, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Χρειάζεται ένα πνεύμα συμβιβασμού και η πολιτική θέληση να εξεύρουμε τις απαραίτητες συμβαστικές λύσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα έχουμε ποτέ μια συμφωνία και από τη δική μας πλευρά το Συμβούλιο θα πράξει όπως και σε όλα τα άλλα συμβούλια θα πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση και τώρα φτάνουμε στην ε, κορονίδα της σημερινής ημέρας κυρίες και κύριοι. θα βγάλουμε φωτογραφίες. Να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Εδώ μπροστά είναι μια